Good afternoon, colleagues. Welcome to Καλησπέρα συνάδελφοι. Καλώ ήρθατε στην απογευματινή μα συνεδρίαση. Πρώτο σημείο στην ημερήσια. Είναι μια παρουσίαση από το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο τη ειδική έκθεση κατά πολέμηση τη πατάλη τροφίμων». Με χαρά λοιπόν καλωσορίζω την κυρία Μπετίνα Γιάκοψεν, και τον κύριο Μάικλ Μπέιν για την ανταλλαγή απόψεων που θα έχουμε μαζί τους. Θα δώσω πρώτο λόγο στον κύριο Γιάκοψεν, μετά θα δώσω το λόγο στα μέλη και θα συζητήσουμε. Καλώ ήρθατε λοιπόν κυρία Γιάκοψεν. Το θέμα σημαντικό για μας, από ό,τι βλέπω και για εσά το ίδιο, μια και κάνατε την έκθεση. Οπότε να ακούσουμε αυτά που έχετε να μας πείτε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία να σας παρουσιάσω σήμερα την ειδική έκθεση του Ελληνικού Συνεδρίου σε σχέση με την καταπολέμηση της πατάλης τροφίμων στην Ένωση. Ήδη είχα παρουσιάσει την έκθεση αυτή σε άλλη επιτροπή, αλλά χάρηκα που, για αλλά χάρηκα που είμαι εδώ σήμερα να την παρουσιάσω και σε εσά σε σχέση με την ε, έκθεση Μποτσάν. Στην ε, σύντομη παρουσίασή μου θα μιλήσουμε για τα ευρήματα της έκθεσής μας και τις συστάσεις της έκθεσης. Όλοι γνωρίζουμε τη σημασία του θέματος της καταπολέμησης της πατάλης τροφίμων. Να σας υπενθυμίσω, σε όλους μας δηλαδή, την οικονομική σημασία αυτού του θέματος, γιατί η σπατάλη τροφίμων είναι ένα θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει όλους τα τελευταία χρόνια και οι υπολογισμοί δείχνουν ότι γύρω στο 1 τρίτο του, των τροφίμων που παράγονται για ανθρώπινη κατανόηση απορρίπτονται ή χάνονται παγκοσμίω. 88 εκατομμύρια τόνοι τροφίμων σπαταλώνται κάθε χρόνο στην Ένωση. Και αυτή η σπατάλη βεβαίω λαμβάνει χώρα σε όλη την διατροφική αλυσίδα κατανάλωση, παρασκευή, κατανάλωση, ε, μεγάλα, μεγάλες επιπτώσεις και για το περιβάλλον. Και τα Ηνωμένα Έθνη υπολογίζουν το κόστος σε πολλά πολλά δισεκατομμύρια ετησίως το χρόνο. Μιλάμε λοιπόν για πολλά χρήματα και αυτή τη στιγμή στην Ένωση δεν έχουμε ορισμό για την σπατάλη τροφίμων. Οπότε δεν είναι δυνατόν να ορίσουμε και να υπολογίσουμε ακριβώς την ποσότητα σπατάλης. Επίσης δεν υπάρχει κοινή βάση μέσω της οποίας θα τεθούν σημαντικοί στόχοι για να γίνουν βελτιώσεις. Όπως ξέρετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως και το Συμβούλιο και η Κομισιόν και ο χώρες μέλη έχουν εκφράσει την επιθυμία τους να καταπολεμήσουν τη σπατάλη των τροφίμων. Και με χαρά είδα ότι το σχέδιο έκθεση τη κυρία Μπόσνας και η δική μα έκθεση είναι ευθυγραμμισμένα ώστε να επιτρέψουμε και στην Κομισιόν να διαδραματίσει πιο σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση τη πατάλη. Μαζί λοιπόν θα πρέπει να του ενθαρρύνουμε ώστε να ενισχύσουν τι δράσει του περαιτέρω στον τομέα αυτό. Στον όλο μα προσπαθήσαμε να δούμε κατά πόσο η Κομισιόν θα μπορούσε να συμβάλλει με μια αποτελεσματική διατροφική αλυσίδα μέσω τη αποτελεσματική καταπολέμησης διατροφική πατάλη. Καταρχά πρέπει να δούμε κατά πόσο η Κομισιόν έχει μεταφράσει τις διάφορες δηλώσεις από δηλώσεις από λόγια σε δράση. Κατά δεύτερο λόγο θα πρέπει να σχεδιαγραφίσουμε τις ευκαιρίες που υπάρχουν για τις κατά πολέμηση της πατάλης που ήδη υπάρχουν σε τωρινές πολιτικές, σε υπάρχουσες πολιτικές. Τι βρήκαμε λοιπόν στην έκθεσή μας. Καταρχά το σημαντικότερο, το γενικότερο μήνυμα της έκθεσης είναι ότι η Κομισιόν δεν καταπολεμά τη σπατάλη, αποτελεσματικά και οι τωρινέ πολιτικέ αλλά και πρωτοβουλίε θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ώστε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο αυτό. Πολλέ πιθανέ βελτιώσει δεν χρειάζονται νέε πρωτοβουλίε ή περισσότερα δημόσια κονδύλια, αλλά απλά μια καλύτερη ευθυγράμμιση των προξών πολιτικών και ένα καλύτερο συντονισμό εντό τη Κομισιόν και μεταξύ Κομισιόν και χωρών μελών. Είδαμε ότι οι δράσει που έχουν λάβει η χώρα μέχρι τώρα ήταν κατακαιρματισμένε και ενα καλυτερο συντονισμο εντο τη κομισιον και μεταξυ κομισιον και χωρων μελων ειδαμε οτι οι δρασει που εχουν λαβει η χωρα μεχρι τωρα ηταν κατακαιρματισμενε και λυπεις και δεν υπάρχει μια πανευρωπαϊκή στρατηγική για την καταπολέμηση τη πατάρη των τροφίμων. Παρά λοιπόν όλο και την, αυξανόμη, την όλο και αυξανόμενη σημασία αυτού του θέματο στο πολιτικό θεματολόγιο, λείπει μια φιλόδοξη στάση. Λείπει ένα κοινό ορισμό και μια επιφανμένη βάση μέσω τη οποία θα αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Υπάρχουν διάφορες πολιτικές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ε, στάση όλων των εμπλεκομένων στη διατροφική αλυσίδα. Παρ' όλα αυτά είδαμε να υπάρχει έλλειψη αποτελεσματική ε, μελέτη αντικτύπου στι πολιτικέ ένωσε σε σχέση με την σπατάλη τροφίμων. Κύριε πολιτικέ όπω η κοινή αγροτική πολιτική, παραδείγματο χάρη, θα μπορούσαν να διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση τη σπατάλη. Και στο πλαίσιο αυτό, λυπάμαι που η Κομισιόν και η Γενική Διεύθυνση Άγκρη δεν είναι διατεθειμένε να αποδεχτούν ότι ο πρωτογενή τομέα και ιδιαίτερα οι γεωργοί έχουν πρωταρχικό ρόλο να διαρματίσουν στην καταπολέμηση τη πατάλη. Και με χαρά είδα λοιπόν ότι η έκθεση της κυρίας, το σχέδιο έκθεση τη κυρία Μπόσαν τονίζει ακριβώ όλε τι δράσει σε όλο το μήκο τη διατροφική αλυσίδα και όχι μόνο στο πλαίσιο των καταναλωτών και των εμπόρων, ώστε να καταπολεμήσουμε δηλαδή την σπατάλη αυτή και η καταπολέμηση αυτή να πάει πέρα αυτών των διαστάσεων. Ένα άλλο που θα ήθελα να τονίσω είναι δωρεά τροφίμων. Κάτι το οποίο είναι πολύ, πολύ αποτελεσματικό τρόπο μείωση τη σπατάλη τροφίμων και το οποίο αναφέρει και το σχέδιο τη κυρία Πόσα. Είδαμε ότι η δωρεά τροφίμων είναι αρκετά περιορισμένη και υπάρχει έλλειψη σαφήνειας και συνοχής όσον αφορά την ερμηνεία των διατάξεων. Τι συστήνουμε λοιπόν από τη δικιά μας την πλευρά. Όπως ήδη ανέφερα, η Κομισιόν έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει όσον αφορά την καταπολέμηση της πατάτη τροφίμων μαζί με τι χώρες μέλη. Η έκθεσή μας περιλαμβάνει διάφορες συστάσεις που θεωρούμε θα μπορούσαν να βοηθήσουν ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική η καταπολέμηση της πατάλης. Καταρχάς, η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την καταπολέμηση θα πρέπει να ενισχυθεί και να, να συντονιστεί καλύτερα. Θα πρέπει η Κομισιόν να χρησιμοποιήσει τα αρχικά βήματα που έχουν γίνει ώστε να αναπτύξει ένα σχέδιο δράση για τα επόμενα χρόνια. Και δεύτερον, μέσω συντονισμού των διαφόρων πολιτικών θα έχουμε περισσότερε δυνατότητε καταπολέμηση. Η Κομισιόν θα πρέπει να λάβει υπόψη τη την σπατάλη στι μελλοντικέ μελέτε αντικτύπου και να θυγαμίσει καλύτερα τι πολιτικέ που καταπολεμούν τη σπατάλη. Και τρίτον, θα πρέπει να διευκολύνουμε την δωρεάν μου που αλλιώ ε, σπατελώνται. Η Κομισιόν μέσω αυτή τη δράση θα μπορούσε να διευκρινίσει παράλληλα και το νομικό καθεστώ που διέπει τι δωρεέ. Θα μπορούσε επίση να θαρρύνει τι περαιτέρω μάλλον περαιτέρω τι υπάρχουσε δυνατότητε για την δωρεά των τροφίμων οικομισιών, ώστε αυτέ να ενταχθούν και σε άλλες πολιτικές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κομισιόν για τη συνεργασία τη σε αυτό τον έλεγχο. και δέσμευση για περαιτέρω βελτιώση. Τώρα, έχει έρθει η ώρα να δείξουμε ότι πραγματικά μιλάμε σοβαρά και ότι Όλε οι πρωτοβουλίε που υπάρχουν, πλατφόρμες, πρωτοβουλίε κτλ. είναι καλέ, αλλά αν δεν έχουμε ένα σαφή ορισμό σπατάλη, αν δεν έχουμε μια σαφή βάση αντιμετώπιση και μια πραγματική και ουσιαστική βούληση ευθυγράμμιση πολιτικών, ώστε να λάβουμε υπόψη μα τον αντίκτυπο αυτή τη σπατάλη, τότε θα έχουμε περισσότερες χαμένες ευκαιρίε στο μέλλον. Και αυτό θα ήταν κρίμα για του Ευρωπαίου πολίτε και για τις μελλοντικέ γενιές που θα πληρώσουν το τίμημα. Τέλος, να ευχαριστήσω την κυρία Μπόσον, την εισηγήτρια της ΕΜΒΗ, επειδή προτίμασε ένα πολύ καλό σχέδιο έκθεσης και θα ήθελα να διατηρήσουμε όλοι μαζί την πίεση προς την Κομισιόν ώστε να δράσει αυτό τον τομέα. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω για τα ερωτήματα που θα έχετε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Λεκύ Πρόεδρος. Μιας και αναφέρεται την κυρία Μπόσαν, να ξέρουμε εσά κύριε Μπόσαν Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Γιάκοψεν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα πολύ ενδιαφέροντα αυτά πράγματα που μας είπατε και βλέπω με χαρά ότι συμφωνούμε σε όλα σχεδόν. Θα ήθελα και εγώ να τονίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι από τις πλέον προηγμένες ε, κοινωνίες ε, στον κόσμο και έχει την ηθική και πολιτική υποχρέωση να περιορίσει τις τεράστιες ποσότητες ε, τροφίμων που απορρίπτονται κάθε χρόνο γιατί αυτό ε, αποτελεί και έλλειψη σε ό,τι αφορά την ε, κατανάλωση πόρων που απαιτούνται για την δημιουργία και την ε, παραγωγή όλων αυτών των τροφίμων, νερό, ενέργεια, πρώτε ύλε, που πολλέ φορέ είναι και περιορισμένοι πόροι. Από το πρόγραμμα Fusion προκύπτει ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση σπαταλούμε περίπου 88 εκατομμύρια τόνους τροφίμων πάνω από 50% αφορά τα νοικοκυριά, 19% τη, τη μεταποίηση, 12% τα εστιατόρια, 10% γεωργία, πρωτογενής τομέας και 5% στο εμπόριο. Όσο συγγήτρια για την ε, έκθεση ε, για την καταπολέμηση ε, της πατάλης τροφίμων, θα θέλω να ευχαριστήσω το ελεκτικό συνέδριο για την εξαιρετική αυτή μελέτη, αυτό το έγγραφο που μας παρουσιάζει και θα ήθελα, έκθεση μάλλον, και θα ήθελα να πω ότι και η χρονική συγκυρία είναι πολύ καλή. Γιατί σε ό,τι αφορά το δικό μας ε, έργο θεωρούμε ότι είναι πολύ επίκαιρη αυτή η συζήτηση. Έχουμε αξιοποιήσει μεγάλο όγκο στοιχείων που προκύπτουν από αυτή την έκθεση και στο δικό μας έργο. Αποτελούν λοιπόν όλα αυτά μια θετική επιρροή ε, στο δικό μας κοινοβουλευτικό έργο. Με την αναθεώρηση θέλουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει σε μια πιο αποδοτική ε, αλυσίδα επιστηστική ε, με τις προσπάθειές της. Και βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν ισχύει κάτι τέτοιο, όμως εντοπίζονται μέθοδοι μέσω των οποίων οι ισχύουσε πολιτικέ μπορούν να εφαρμοστούν πιο αποτελεσματικά για να καταπολύσουμε το πρόβλημα. Το Ελεκτικό Συνέδριο επίση έχει ε, αναφέρει ότι για πολλέ από αυτέ τι βελτιώσει που αναφέρει η κυρία Γιάκοψεν δεν χρειαζόμαστε νέε πρωτοβουλίε ή ε, αυξημένη χρηματοδότηση. Χρειαζόμαστε μια καλύτερη ευθυγράμμιση ε, των υπαρχουσών πολιτικών, καλύτερο συντονισμό και πιο σαφή μέτρα για την αποτροπή σπατάλης τροφίμων. Και παρόλη την αυξανόμενη ε, σημασία αυτών των προγραμμάτων, το Ελληνικό Συνέδριο κρίνει ότι το επίπεδο φιλοδοξίας ε, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια. Θεωρούν επίσης ότι είναι κατακαιρματισμένα, ελλειπή και λοιπόν συντονισμένα τα μέτρα από πλευρά τη Κομισιόν. Σε ό,τι αφορά τι ε, δωρεέ φαγητών, ε, υπάρχουν για παράδειγμα διαφορετικέ ερμηνείε τη ισχύουσα νομοθεσία και αυτό, τέτοιου τέτοια είδου προσκόμματα μπορούν να αρθούν προκειμένου οι δωρεέ τροφίμων να ε, απλουστευτούν για να αποφύγουμε τη σπατάλη. Γιατί όμως έχουμε τέτοια τεράστια σπατάλη φαγητού και τροφίμων. Είναι σύνθετη η απάντηση και πολύ επίπεδη. Πολλέ φορές οι ίδιοι αγρότε δεν μπορούν να πουλήσουν το εμπόρευμά του και το αφήνουν να σαπίζει στα χωράφια. Ε, οι μεταποιητές κάποιες φορές ε, αξιοποιούν μόνο τμήμα τη πρώτη ύλη και, ε, και πετούν το υπόλοιπο. Και οι έμποροι κάποιες φορές μπορούν να μην το πουλήσουν, είναι δύσκολοι αυτούς να το δωρήσουν και έτσι το πετούν. Και οι καταναλωτέ, βέβαια πολλές φορές σπαταλούν το φαγητό. Σε όλα αυτά τα στάδια λοιπόν βλέπουμε πώς μπορούμε να περιορίσουμε τη σπατάλη ή να αυξήσουμε τη δωρεά των τροφίμων ε, είτε για την ανθρώπινη κατανάλωση είτε και για άλλες μορφές όπως είναι ε, η κομποστοποίηση. Είναι λοιπόν σύνθετο το ζήτημα, γι' αυτό χρειαζόμαστε μια συντονισμένη πολιτική σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο και εκεί θα πρέπει να εμπλέκονται όλοι οι ενδιαφερομενοί φορείς. Αυτή τη στιγμή έχουμε 52 ε, κανονιστικές ε, διατάξεις που ε, διέπουν τη σπατάλη τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 29 είναι κανονισμοί, 10 οδηγίες, 3 αποφάσεις και 10 συστάσεις. Πρόκειται λοιπόν για νομοθετικές τάξεις, πράξεις από τον τομέα του περιβάλλοντος, της υγείας, ε, προστασία καταναλωτών, περιβάλλοντος και εμπορίου. Η έκθεση την οποία εκπονώ θα θίξει πολλέ από αυτές τις πτυχέ και θα εντοπίσει και του τομείς που, όπου δεν υπάρχει επαρκής ρύθμιση και όπου ε, η εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών μπορεί να επωφελήσει ε, την πολιτική μας αυτή. Στις τροπολογίες που έχω συντάξει αναφέρουμε ότι οι καταναλωτές πολλές φορές επομίζονται το βάρος ε, της πατάλης τροφίμων και τα κράτη-μέλη δεν αξιοποιούν το, ε, τα προγράμματα για το γάλα και τα φρούτα στο σχολείο και ότι δεν κάνουν αρκετά ε, για να καταπολεμήσουν τις πρακτικέ πρακτικές ε, στο εμπόριο. Η έκθεση θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμπεριλάβει την ε, σπατάλη τροφίμων στην νομική ανάλυση αντικτύπου και να δούμε τον αντίκτυπο της κοινή γεωργικής πολιτικής και της κοινή αλληλευτική πολιτικής. Πρέπει να γίνει καλύτερη χρήση των διαθέσιμων πόρων, ιδιαίτερα για τους πλέον μειονεκτούντες του ταμείου αυτού δηλαδή, ε, να, και να αυξηθούν οι δωρεές τροφίμων. Θα αναφερθούμε και στο μεγαλύτερο τμήμα των συστάσεων του Λεπτικού Συνεδρίου. Ε, εγώ προσωπικά συμφωνώ με αυτή την ε, συνέργεια, δηλαδή την κοινή πίεση μπορούμε να ασχίσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κρατημέλη. Σας συγχαίρω και πάλι λοιπόν για την έκθεσή σας. Συγχαίρω την ομάδα του Ελληνικού Συνεδρίου, τη οποία ηγήθηκε η κυρία Γιάκοψεν, ε, για ένα πολύ χρήσιμο και επίκαιρο ζήτημα και κείμενο. Ευχαριστούμε πολύ, λέει Πρόεδρο. Κυρία Δελάκη. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κυρία Ντελαέ, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω το Ελληνικό Συνέδριο για αυτή την μελέτη, η οποία πραγματικά είναι ιδιαίτερα επίκαιρη. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια διαδικασία στοχασμού και προβληματισμού Όλοι θα συμφωνήσουμε απολύτως με τα όσα μας είπατε, όμως έχω κάποιες διαφορετικές ε, σκέψεις. Το βασικό για μας ε, είναι να ξαναδώσουμε την σημασία και την αξία που έχουν αυτά τα τρόφιμα. Γιατί όταν τα πετάμε είναι σαν να λέμε ότι αυτά τα τρόφιμα δεν είναι αγαθά και ότι δεν έχουν αξία. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε και τους πολίτες. Θα πρέπει λοιπόν ε, ε, να διεξαγάγουμε εκστρατείες, ε, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κατά της πατάλης τροφίμων, κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Μεταξύ άλλων μιλήσατε και για τον πρωτογενή τομέα, όχι μόνο για αυτόν βέβαια. Εγώ αυτό που δεν άκουσα είναι η διαφορά μεταξύ των απολειών και της σπατάλης. Στο στάδιο της παραγωγής είναι σημαντικό αυτό το μερίδιο. Γιατί έτσι δίνουμε την εντύπωση ότι οι γεωργοί απλώς σπαταλούν έτσι χωρίς λόγο. Εγώ είμαι γεωργός και μπορώ να σας πω ότι η μοναδική μου βούληση είναι να θρέψω του συμπολίτε μου, όχι να πετάξω τρόφιμα χωρίς λόγο. Υπάρχουν κάποιοι λόγοι όμω ε, ε, για, για αυτές τις απώλειες. Εγώ εδώ και μερικά χρόνια ε, δημιούργησα μία ένωση ε, που κάνει ακριβώς αυτό που ε, προκειμένου τα τρόφιμα που δεν μπορούν να πωλήσουν οι γεωργοί να μπορούν να τα διαθέσουν στους συμπολίτες μας που δεν έχουν τρόπο να τραφούν σωστά. Και κάτι τελευταίο, μιλήσατε για την ε, συνοχή των ευρωπαϊκών και συνάφεια των ευρωπαϊκών πολιτικών. Πολύ σωστό, όμω δεν πρέπει να ζητούμε από την κοινή γεωργική πολιτική να ρυθμίσει πράγματα για τα οποία δεν έχει δημιουργηθεί. Δεν είναι αυτό ο σκοπό. Βεβαίω θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, και αυτή την προβληματική, όμω από την άλλη το να γίνει στόχο αυτό για την κοινή γεωργική πολιτική νομίζω ότι εκεί είναι λάθο η μάχη που επιλέγουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Λεκή Πρόεδρος. Σκρελέκ τώρα. Παρακαλώ κύριε Σκρελέκ. Ο Σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Επιτρέψτε μου καταρχάς εκ μέρους των Πρασίνων να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στο ελεκτικό συνέδριο για μια εξαιρετική έκθεση. Είμαι ο εισηγητής ε, που ε, ασχολείται με το πακέτο της κυκλικής οικονομίας και το θέμα αυτό είναι κάτι που μας έχει απασχολήσει και έχουμε δουλέψει πάνω σε αυτό αρκετά. Γι' αυτό θεωρώ πως είναι αναγκαίο η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι αποτελεσματική στην προσπάθεια καταπολέμησης της πατάλης τροφίμων. Αυτό που ακούσαμε σήμερα και από την εισηγήτρια και από το ελεκτικό συνέδριο ε, δείχνει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εργάζεται αποτελεσματικά. Γι' αυτό θα ήθελα να καλέσω και την Επιτροπή και τα κρατημέλη να προσπαθήσουν να καταπολεμήσουν πραγματικά τις σπατάλη τροφίμων. Και Λυπάμαι πολύ για το ότι οι συνάδελφοι ευρωβουλευτές δεν είναι ιδιαίτερα ενεργοί στις ε, προσπάθειές τους καταπολέμησης αυτής της πατάλης πέρα από τα προβλήματα στην νομοθεσία, πολλές φορές ακούμε ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα, περισσότερα να αυξηθεί η παραγωγή τροφίμων, ε, ακούμε για τους ε, γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, αλλά πρέπει να κοιτάξουμε την υγεία των πολιτών. Αυτό είναι το κύριο μέλημά μας και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κάνουμε αντιφατικέ ενέργειες που θα οδηγήσουν στη σπατάλη τροφίμων. Είναι επίσης και ένα πρόβλημα δεοντολογίας, ηθικής αν θέλετε. Μπορούμε να το δούμε και από αυτή τη σκοπιά. Ε, με τα χαράς λοιπόν να ενσκύψω πάνω σε αυτό το θέμα της πατάλης τροφίμων στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας. Ορισμένοι ίσως θεωρούν πως δεν χρειάζεται ορισμός αυτού ε, του όρου, αλλά εγώ πιστεύω πως πρέπει να γίνει κάτι. Καταρχάς πρέπει να προσδιορίσουμε το πρόβλημα, να το ορίσουμε, να το περιγράψουμε. Και θα ήθελα τέλος να κάνω και μία ερώτηση στους εκπροσώπους του Ελεκτικού Συνεδρίου. Εσείς έχετε κάποιες συστάσεις προς τους ευρωβουλευτές. Μπορείτε να μας πείτε τις δικές σας ιδέες για το πώς μπορούμε να ανεβάσουμε αυτό το θέμα στη λίστα των προτεραιοτήτων. Σας ευχαριστώ πολύ. Η ε, κυρία Ζόμερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμότατα το Ελεκτικό Συνέδριο για αυτήν την έκθεση. Είναι ένα πρόβλημα πραγματικά πολύπλοκο και πολυδιάστατο η σπατάλη τροφίμων και πιστεύω πως το πρόβλημα αρχίζει ακριβώς από ε, το σημείο του ορισμού. Δεν έχουμε κάποιον ακριβή ορισμό για αυτό το θέμα, το ανέφεραν ήδη και άλλοι συνάδελφοι και αναφέρθηκαν επίση στο ε, ερώτημα του τι είναι απώλεια, τι είναι σπατάλη υπάρχουν τρόφιμα που πετιούνται, που σπαταλούνται και αυτό είναι και απώλεια εισοδήματο για ορισμένους. Υπάρχει επίσης και απώλεια στη εισοδιά των αγροτών, αλλά αναρωτιέμαι και αν αυτή η ζημιά, η καταστροφή της οδιάς ε, προέρχεται και από ε, άλλους παράγοντες. Αν, πούμε, για παράδειγμα, συνυπολογίζονται και τα διάφορα ε, ζυζάνια και οι διάφορες ε, ασθένειες των ε, φυτών. Ε, δηλαδή εάν το πρόβλημα εντοπίζεται και στην πρωτογενή παραγωγή. Επίσης, θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτό που άκουσα πριν, ότι σίγουρα δεν είναι υπεύθυνο μόνο το εμπόριο και τα νοικοκυριά, αλλά πρέπει να παραδεχτούμε ότι το 35% της σπατάλης τροφίμων ε, οφείλεται ακριβώς σε αυτά τα νοικοκυριά, στον καθένα μας δηλαδή. Ε, είναι πρόβλημα και αυτό είναι κάτι που ε, συζητούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, το ότι δηλαδή ο κόσμος ελάχιστα πράγματα γνωρίζει για τα τρόφιμα, τι ακριβώς είναι, ε, πώς δημιουργούνται. Ο κόσμος μπορεί να γνωρίζει, την, μπορεί να γνωρίζει πολλά και να βλέπει πολλά τρόφιμα στα σούπερ μάρκετ, αλλά δεν είναι ενημερωμένος, δεν ξέρει πώς μπορεί να μαγειρέψει για παράδειγμα κάτι και αυτό οδηγεί σε άλλα προβλήματα για παράδειγμα, ε, την ε, αύξηση των ποσοστών παχυσαρκίας στον πληθυσμό. Ε, επαναλαμβάνω, τα κράτη-μέλη βρίσκονταν σε λίθαργο, τα, τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, τα ασφαλιστικά συστήματα βρίσκονται σε λίθαργο. Δεν αναγνωρίζεται παρκώς η αξία των τροφίμων. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, διότι πρέπει καταρχάς να ξέρουμε πόσο μεγάλη είναι η αξία αυτού που θα καταναλώσουμε για να μπορέσουμε να το εκτιμήσουμε. Ε, τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Η γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού επίσης. Το 80% του πληθυσμού της Ευρώπης ζει στις πόλεις και από εκεί αρχίζει το πρόβλημα. Υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης στα σχολεία, υπάρχει απομάκρυνση του κόσμου από, ε, από την ίδια την παραγωγή, από το τρόφιμο. Γι' αυτό πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα εκεί. Ενημέρωση, παιδεία. Και η έλλειψη επαρκούς παιδείας πιστεύω πως είναι ένα οφθαλμοφανές φαινόμενο. Χρειάζεται λοιπόν η ενημέρωση, η γνώση για όλον τον κύκλο των τροφίμων να, ε, να γίνει κτήμα όλο ένα και περισσότερων πολιτών. Επίσης πρέπει να υπάρχει επαρκή ενημέρωση για την ημερομηνία λήξης ενός προϊόντος που πολλές φορές ε, δεν σημαίνει ότι με το που ε, παρέλθει αυτή η ημερομηνία πρέπει να το πετάξουμε. Πολλέ φορέ διαβάζει κάποιο την ημερομηνία, βλέπει την ημερομηνία λήξη, λέει Αχ, χθεσινό, το πετάω. Ενώ στην πραγματικότητα διαφέρουν πολύ τα πράγματα, είναι ε, δυνατόν να το καταναλώσει κάποιο. τώρα, Σίγουρα οι βέλτιστε πρακτικέ και η ανταλλαγή αυτών από τα κράτη-μέλη θα βοηθήσει, αλλά δεν ξέρω αν είναι ανάγκη να δημιουργήσουμε μία καινούργια πλατφόρμα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους ε, ήδη υφιστάμενους ε, πόρους που διαθέτουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, δεν είδατε που μόλι περάσαν τα δύο λεπτά σας κανένα νόημα. Πρέπει να τηρήσουμε το, τους χρόνους ομιλίας. Λοιπόν, α προχωρήσουμε. Κλείνω και τον κατάλογο των ομιλητών. Η κυρία Κρούπα έχει το λόγο. Δύο λεπτά έχετε. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Όπως ακούσαμε και όπως ε, συζητάμε, ένας από τους ε, πολλούς λόγους της σπατάλης ε, τροφίμων είναι η αξία των τροφίμων. Η αξία των τροφίμων υποβαθμίζεται όλο ένα και περισσότερο. Στην Πολωνία υπάρχουν, από όσο ξέρω, σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία ενημερώνουν τους πολίτες ότι ναι, δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις για παράδειγμα κάποια κομμάτια του κοτόπουλου γιατί έχουν ε, αντιβιωτικά, είναι γεμάτα κολαγόνο, τα λαχανικά έχουν φυτοφάρμακα σε αυτό και σε αυτό το κομμάτι τους, ενημερώνονται για τα πρόσθετα, για τα διαφορετικά φυτοφάρμακα λοιπάσματα που χρησιμοποιούνται, γίνεται κάτι. Αυτό όσον αφορά τις βέλτιστες πρακτικές. Μετά, να σας πω επίσης πως ε, πρόσφατα στην Πολωνία έγινε θέμα, το, θέμα, ε, το ζήτημα της παραποίησης τροφίμων. Υπάρχουν, ξέρετε πολλοί που κάνουν μια περιουσία με αυτές τις περίεργες σκοτεινές δραστηριότητες. Και αυτό με φέρνει στο επόμενο θέμα που ήθελα να θίξω, τις κυρώσεις. Υπάρχει έλλειψη ελέγχων και οι κυρώσεις δεν είναι τόσο αυστηρές όσο θα έπρεπε. Γι' αυτό λοιπόν Αναρωτιέμαι εάν είμαστε υπερβολικά χαλαροί με την νομοθεσία, αν υπάρχει υπερβολική έλλειψη ελέγχου. Στην Πολωνία μα λένε ότι πρέπει να υπάρχουν ετικέτες στα πάντα, να υπάρχει ένας πλήρης κατάλογος των συστατικών. Τη δεκαετία του 90 άρχισαν οι πρώτες προσπάθειες αυτές, αυτής της ε, παραποίησης, της, ε, της τροφίμων. Ήδη από τότε, ήδη τότε βρίσκουμε τις ρίζες. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι το θέμα της αξίας των τροφίμων πρέπει να αντιμετωπιστεί καταρχάς ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. τώρα, οι αγρότες δεν παίρνουν παρά ελάχιστα χρήματα για τα προϊόντα τους και τα σούπερ μάρκετ αντίθετα κερδίζουν πολλαπλάσια. Χρειάζεται λοιπόν η θέσπιση κάποιων κανόνων για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό. Τώρα δεν θα αναφερθώ στα υπόλοιπα, αλλά θα τα διαβάσετε στις τροπολογίες μου. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φλόρεντς. Ε, με όλο το σεβασμό προς την συνάδελφο ιατρό στην Πολωνία, ε, πρέπει να φέρω κάποιες αντιρρήσεις. Πιστεύω ότι εσείς μπορείτε να αλλάξετε τα πράγματα. Δεν πρέπει να ζητάτε νομοθεσία από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να προστατεύσετε ε, τους πολίτες. Η ίδια η κυβέρνησή σας τι κάνει. Μετά, καταρχάς, να ευχαριστήσω την εκπρόσωπο του Ελεκτικού Συνεδρίου για την έκθεση και επιτρέψτε μου να βάλω έτσι λίγο χιούμορ στην κουβέντα μας. Μέχρι την τελευταία κοινοβουλευτική θητεία η Επιτροπή Περιβάλλοντος ήταν η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή σε αυτό το θέμα. Υπήρχε μάλιστα μία ε, υψηλά ιστάμενη κυρία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία τράβηξε μία χοντρή κόκκινη γραμμή και μας είπε μέχρι εδώ. Φτάνει. Περνάει το θέμα στη Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ. Και έκτοτε άλλαξαν τα δεδομένα, δεν λαμβάνεται υπόψη η άποψη της Επιτροπής μας και γενικά δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει. Εσείς τι πληροφορίες έχετε για αυτά που έχουν γίνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα, να πω πως οι δύο συνάδελφοι από την πολιτική μου ομάδα μίλησαν για τη σπατάλη μόνο. Εγώ δεν έχω να προσθέσω πάρα πολλά σε αυτό θα ήθελα μόνο να πω ότι όταν πηγαίνω στο μανάβι, ας πούμε στο σούπερ μάρκετ να αγοράσω πατάτες, ε, τα πάντα είναι, σχεδόν τα πάντα είναι από την εταιρεία McCain. Και τι μου είπαν ότι εάν ας πούμε οι πατάτες, μου είπαν οι αγρότες που προμηθεύουν τη McCain, ότι αν οι πατάτες δεν έχουν ένα συγκεκριμένο μέγεθος, τις πετάνε. Αν δεν, είναι, ε, αν δεν έχουν διάμετρο τουλάχιστον 3 εκατοστά. Στα σκουπίδια. Και το ίδιο συμβαίνει και με τα σαχαρότεφλια. Και το θέμα δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι ότι πετάμε τα τρόφιμα. Το θέμα είναι ότι υπάρχει και πρόσθετο κόστος για την συγκομιδή αυτών των απορριμμάτων. Εντό εισαγωγικών απορριμμάτων. Και ε, αυτό είναι το πρόβλημα. Ε, αρχίζουμε από αυτές τις μεγάλες πολυεθνικές, τη Μακέι, να πάμε και στα McDonald's που μας κάνουν τη ζωή δύσκολη με αυτές τις πρακτικές τους. Και ξέρετε, ένα μικρό μαυράκι να υπάρχει πάνω στην πατάτα, ένα μικρό ματάτι, ε, μαυράκι, το οποίο δεν φαίνεται όταν πλύνεις την πατάτα, ε, το πετάνε. Χαλάει την εικόνα. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε σύντομοι παρακαλώ. Θα ήθελα να πω στους συναδέλφους ότι στην Πολωνία ένα μεγάλο ποσοστό, κοντά στα 50% των τροφίμων, έρχεται από το εξωτερικό. Ναι, λέει ο κύριο Φλόρεντ, αλλά τι έλεγχοι γίνονται στη χώρα σα. Αυτό είναι το θέμα. Εσεί τι πιστεύετε. Είναι μια πολύ χρήσιμη η σημερινή συζήτηση. Θα ήθελα πρώτα να πω αυτό που ανέφερε ο κύριος Φλόρενς ε, μόλις τώρα και η κυρία Σόμερ, αλλά και η κυρία Ντελέ, η σχεδόν της Ό,τι αφορά τη Γεωργία, Είναι ε, πολύ σημαντικό το ζήτημα της, ε, του καθορισμού της τιμής με βάση την ε, ζήτηση. Ε, δεν χρειάζεται εμείς να ασχοληθούμε με όλο αυτό, γιατί πολύ μεγάλο κομμάτι των απολειών χρησιμοποιείται ω ζωοτροφή από τους Γιώργους. Υπάρχει ορκνομοθεσία λοιπόν και στη χώρα μου και ευρύτερα. Και το δεύτερο είναι ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ε, αυτά τα απορρίμματα ε, σε ειδικέ εγκαταστάσεις ε, ως μορφή ενέργειας. Πρώτα απ' όλα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στους ανθρώπους και να τους ενημερώσουμε. Και στο σχολείο μάθαμε πράγματα για τα τρόφιμα και την τροφή, όμως από εκεί και πέρα τι θα κάνουμε. Πρέπει να ενημερώσουμε και τους καταναλωτές τι αγοράζουν και γιατί και με τον κύριο Ντροσκάτη τα έχουμε συζητήσει όλα αυτά. Πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό και κλείνοντα. Σε ό,τι αφορά τον κλάδο του επιστημισμού, να πω ότι μπορούν όλοι, για παράδειγμα, να μικρύνουν τις μερίδες και έτσι να είναι λιγότερα τα απορρίμματα. Ας μην ασχοληθούμε λοιπόν με τα πάντα στην Ευρώπη, ας μείνουμε στα πιο βασικά. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μιλιό. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ήδη αναφέρθηκαν πολλοί από τους συναδέλφους που ήθελα να πω και εγώ. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω θερμότατα την κυρία Γιάκοψεν για την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. Πιστεύω πως ήταν ιδιαίτερα σημαντικό να έχουμε αυτή την έκθεση ε, γιατί διαβάσαμε πολλά σημαντικά πράγματα. Να ευχαριστήσω επίσης και την εισηγήτρια την κυρία Μπόζαν. Κατά τη συζήτησή μας νομίζω πως ξεχάσαμε το ότι κατά τη διάρκεια παρασκευής τροφίμων ε, σπαταλώνται και ενεργειακοί πόροι αλλά και εκλείται διοξιδίου του άνθρακα. Και αυτό πρέπει να το συνυπολογίσουμε στην σπατάλη των ίδιων των ε, τροφίμων και όπως γνωρίζετε Υπάρχει τώρα νομοθετικά η εντολή, το ίμιση των ε, τροφίμων που πετιούνται να προσπαθούμε να το διατηρήσουμε. Το κάνουν και σούπερ μάρκετ και πολλά. Ε, τι γίνεται με αυτό. Οι συνάδελφοί μου το ανέφεραν επίσης πως πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός ανάμεσα στην απώλεια και τη σπατάλη και να δοθεί ένας ορισμός και των δύο. Τι εννοούμε ε, με τον όρο απώλεια. Πολλές φορές η απώλεια είναι σπατάλη. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν ε, αποθηκεύονται τα τρόφιμα σε κατάλληλες συνθήκες και χαλάνε, αυτό δεν είναι απώλεια, είναι σπατάλη. Και ας δούμε τώρα τι γίνεται και στα κράτη-μέλη. Στη Γαλλία, ας πούμε, υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές, υπάρχουν νόμοι ε, που περιγράφουν τι ακριβώς πρέπει να γίνεται με τα τρόφιμα, τι ακριβώς πρέπει να κάνουν τα σούπερ μάρκετ, τι ακριβώς πρέπει να κάνουν εταιρείε catering. Αυτή τη στιγμή η Γαλλία είναι πρωτοπόρο. Στην ε, Γερμανία, στο Βερολίνο, Υπάρχει μια άλλη πρωτοβουλία που έχουν αναλάβει ε, ορισμένα εστιατόρια. Για παράδειγμα, όσε μερίδε φαγητού στο τέλο τη ημέρα ε, δεν έχουν καταναλωθεί, δίδονται σε άτομα που έχουν ανάγκη. Αυτά πιστεύω είναι πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε, να δούμε πώς μπορούμε να ανταλλάξουμε βέλτιες πρακτικές κτλ. Τέλος, η ημερομηνία λήξης ε, δεν είναι το ίδιο με την ε, ημερομηνία ε, κατανάλωσης. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ντάλη έχει το λόγο. Thanks a lot. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να ευχαριστήσω κυρίως την κυρία Γιάκοψεν για αυτή την σημαντική συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Μπόζαν επίσης που έκανε πολύ καλή δουλειά με την έκθεση. Και το λέω αυτό επειδή εδώ έχουμε ένα πολύ καλό παράδειγμα το πώς τα δύο θεσμικά όργανα μπορούν να συνεργαστούν ώστε να δώσουμε έμφαση σε αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα και ιδιαίτερα, όπως λέει και η Μπιλιάνα, επειδή το θέμα αυτό δεν είναι μόνο πολιτικό αλλά και θέμα ηθικής και είναι πολύ ανησυχητικό βλέποντας τα στοιχεία της έκθεσής σας. Και λάβουμε υπόψη μας το ότι ο κάθε Ευρωπαίος σπαταλάει 180 κιλά κάθε χρόνο. Δεν είναι καθόλου αστείο λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό πόρος. Επίσης στην έκθεσή σας λέτε ότι η Κομισιόν δεν καταπολεμά αποτελεσματικά την σπατάλη και λέτε ότι οι φιλοδοξίες δεν επαρκούν. Αλλά αυτό μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον ότι δεν θέλετε νέε πρωτοβουλίε, αλλά σωστή εφαρμογή των πρωτοβουλίων που ήδη υπάρχουν. Αφερθήκατε σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα στην ανάγκη για μελέτες αντικτύπου όσον αφορά τι πρωτοβουλίε πολέμηση. Θα ήθελα λιγάκι να το αναπτύξετε αυτό, να μας πείτε συγκεκριμένα πώς οι μελέτες αντικτύπου θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν σε επίπεδο πολιτικής. Ακούσαμε για τα διάφορα αγροτικά θέματα, αλλά θα ήθελα τη δική σας άποψη. Το πώς μπορούμε να κατευθύνουμε τις γεωργικές πολιτικές, ώστε να έχουμε χαμηλότερη σπατάλη διατροφικών προϊόντων. Αλλά εκτός από τα θέματα πολιτικής, Τι γίνεται με τη σπατάλη των οικοκυριών και το πώς θα μπορούσαμε να προωθήσουμε την ευαισθητοποίηση για αυτή τη μεγάλη πρόκληση και κάτι άλλο. Δωρεά τροφίμων που αναφέρατε και εσείς και η κυρία Μπόρζαν. Αναφερθήκατε στην απάλληψη στοιχείων αποτροπής δωρεάς, αλλά μέσω ποιων μέτρων μπορεί να γίνει αυτό, ώστε να προωθήσουμε την δωρεά τροφίμων και να μας βοηθήσει αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πατητσίνη. Πρώτα ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ το Ελεκτικό Συνεδρίο για την έκθεση αυτή, για την αντιμετώπιση της πατάλης. Εμείς εδώ ήδη το έχουμε αντιμετωπίσει αυτό το θέμα στα πλαίσια της κυκλικής για τα απορρίμματα. Αλλά και στην δικιά μας πρωτο... έκθεση πρωτοβουλία για τα απορρίμματα τροφίμων. Είναι αλήθεια ότι πριν το 2025 θέλαμε μια μείωση 35% και ανάλογα στη συνέχεια. Είναι όμως σαφές ότι για μας έχει δίτερο ρόλο η πρόληψη. Ο κύριος στόχος μας είναι το να επενδύσουμε στα προγράμματα ενημέρωσης, κυρίως στα σχολεία και σε μια καλύτερη ενημέρωση των ε, πολιτών ώστε να προλάβουμε την σπατάλη, ακολουθώντα την ιεραρχία που υπάρχει. Δίνοντας έμφαση στα τρόφιμα τα οποία προέρχονται για ανθρώπινη κατανάλωση και μετά αυτά για ζωική κατανάλωση. Αλλά επίσης είπαμε κάτι και για τα οργανικά απόβλητα. Θέλουμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται με τα προϊόντα τα οποία δεν πολλούνται και να προωθήσουμε και την δωρεά. Ερώτημα. Κατά την έποψή σας αυτά τα μέτρα επαρκούν για να πετύχουμε τους στόχους οι οποίοι έχουν ε, ενταχθεί στα δικά μας τα έγγραφα και τις εκθέσεις που έχουμε εκπαιδεύσει μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τελειώσαμε με τον κατάλογο των ομιλητών. Θα καλέσω τώρα τον κύριο Γκρούμπαλ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία να απαντήσω σύντομα και να παρουσιάσω την βούληση της Κομισιόν και τη δέσμευσή της για την αντιμετώπιση της σπατάλης. Θα ήθελα να διασκεδάσω ανησυχίε και του ελεκτικού συνεδρίου αλλά και των μελών της Επιτροπής σας ότι δεν έχουμε δέσμευση και βούληση για αυτό το θέμα. Εμείς εδώ συνειδητοποιούμε ότι έχουμε να κάνουμε με ένα οριζόντιο ζήτημα το οποίο αφορά πολλές ε, πολιτικές Υπάρχουν πολλά ωφέλη τη καταπολέμηση τη πατάλη, αυτά είναι προφανή, μέσω καλύτερη βέβαια διαχείριση των πόρων και μιλήσαμε για την γεωργία και πόρου εκεί, αλλά και στον τομέα τη αλληλεία επίση. Μαζί με τι επιπτώσει για το περιβάλλον, παραγωγικότητα κτλ. Αυτά τα έχουμε συνειδητοποιήσει, όπω επίση και τη δυνατότητα χρήση τροφίμων για να στηριχτούν οι ασθενέστεροι. Έχουμε λοιπόν δέσμευση για την επίτευξη περαιτέρων στόχων, ώστε να έχουμε μια συνολική προσέγγιση που θα αφορά όλες τις πολιτικές μας. Έχουμε και ένα σχέδιο δράσης που έχουμε χαράξει στα πλαίσια τη κυκλική οικονομία και η Γενική Διευθυνσία ΣΑΝΤΕ μαζί με τι υπόλοιπε υπηρεσίες τη Κομισιόν και όλου του παρόντε εδώ νομίζω ότι είναι αφοσιωμένοι προσυλλομένοι στους στόχου αυτού. Οπότε δεν υπάρχουν λόγια ανησυχία. Βέβαια χρειαζόμαστε και την δέσμευση όλων των εμπλεκομένων και των χωρομελών αλλά και των φορέων της διατροφική αλυσίδας, δηλαδή ξεκινώντας από την παραγωγή και καταλήγοντας στους καταναλωτές. Έχουμε και μια νέα πλατφόρμα, την οποία αναφέραν διάφορα μέλη τη Επιτροπή σας, Τώρα να δούμε κατά πόσο αυτή η πλατφόρμα είναι σωστό εργαλείο για να πετύχουμε τους στόχους για την πρόληψη και αποτροπή της πατάλης. Εμείς πάντως την ε, προσθέμενη αξία που βλέπουμε σε αυτό το εργαλείο είναι ότι επιτρέπει την ανταλλαγή πρακτικών και την εμπλοκή όλο και περισσότερων φορέων Η δουλειά που έχει γίνει μέχρι τώρα στις πρώτες ανταλλαγές στα πλαίσια αυτού φόρουμ ήταν πολύ καρποφόρες και είναι πολλά υποσχόμενες για τις συζητήσεις που έχουμε προγραμματίσει αργότερα μέσα στο έτος. Το σχέδιο δράσης τώρα που έχουμε παραβάλλει βεβαίως πολλά παραδοτέα τα οποία αφορούν θέματα τα οποία ανέφεραν εδώ και τα μέλη τη Επιτροπής και που έκανε έκκληση για δράση. Δηλαδή περιγράφουμε ας πούμε τι αποτελεί σπατάλη. Α πούμε φέτος ε, θέλουμε να έχουμε ένα ορισμό τη σπατάλη και βεβαίω θα έχουμε μελλοντικά ανταλλαγές απόψεων σε σχέση με την οδηγία πλαίσιο κάτι το οποίο θα αποτελέσει ευκαιρία για όλα τα θεσμικά όργανα να συζητήσουν αυτό το ζήτημα. Πάντω, εμεί από τώρα εργαζόμαστε πάνω σε μια μεθοδολογία ώστε να έχουμε μια συγκεκριμένη περιγραφή και γι' αυτό ακριβώ δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε ω Κομισιόν νομική περιγραφή, αλλά μια ξεκάθαρη τωρινή περιγραφή σε όλη τη διάρκεια τη αλυσίδα, δηλαδή τι αποτελεί σπατάλη και αυτό να αποτελεί τέλο πάντων τη βάση δράση και χάραξη στόχων. Σα ε, βεβαιώ ότι αυτή η στόχη δεν είναι 30% μόνο, είναι 50% ή παραπάνω από αυτό που αναφέρθηκε προηγουμένω. Βεβαίω θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη εποπτεία της ε, σπατάλη τροφίμων. Άκουσα και αυτά που είπατε και τις εκκλήσεις για την δωρεά τροφίμων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό επίση. Έχουμε ένα νομικό πλαίσιο το οποίο όμω ερμηνεύεται τρόπο στι χώρε μέλη από τι αρμόδιε αρχέ. Και ήδη οι εμπλεκόμενοι το εκλαμβάνουν διαφορετικά. Σε σχέση δηλαδή με το δυναμικό της δωρεάς τροφίμων. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο εμείς εργαζόμαστε πάνω σε κάποιες κατευθυντήρες γραμμές για τη δωρεάν τροφέμων. Και το θέμα του μπειτή e που ακούστηκε προηγουμένως στη συζήτηση ώστε να υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα για το θέμα αυτό και λαμβάνουμε υπόψη μας και την έκκληση που προέρχεται από εσά στα πλαίσια ενός πολιτικού προγράμματος για την διάχυση των πρακτικών και της γνώσης που υπάρχει σε αυτό το θέμα, ώστε να βοηθηθούμε περισσότερο. Επίσης σημαντικό είναι και άλλο στοιχείο που ακούσαμε μέσα στη συζήτηση και που αφορά την σύσταση που έκανε η Κομισιόν και που ήδη έχουμε προχωρήσει. Νομίζω ότι συμφωνούμε επίσης για τις πιθανές επιπτώσεις των τωρινών πρακτικών, για τη σημασία της ε, συνειδητοποίησης των καταναλωτών για τη σημασία του θέματος αυτού, όλων των εμπλεκομένων, ε, επισήμανση, ημερομηνία λήξης, ώστε να έχουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία στη διάθεσή μα και να μα βοηθήσουν να πάρουμε σοβαρέ πολιτικέ αποφάσει στο μέλλον. Όλα αυτά λοιπόν τα κάνουμε στην Κομισιόν ώστε πραγματικά να καταλάβουμε ακριβώ τι γίνεται όλοι μα και εμεί ω Κομισιόν και οι εμπλεκόμενοι και οι αρμόδιε αρχέ. Και βεβαίω δεν παραβλέπουμε το ότι όλε οι δραστηριότητε σε αυτό το τομέα δεν θέτουν αμφιβόλο είναι την δέσμευσή μα για υψηλή ασφάλεια στα τρόφιμα και βεβαίω υπάρχουν και άλλα εργαλεία για την διασφάλιση αυτής της ποιότητας των τροφίμων. Θα θυμάστε, Πρόεδρε, την πρόσφατη συμφωνία και την πρόταση της Κομισιόν για τους επίσημους ελέγχους που θεωρούμε ότι είναι πολύ καλά εργαλεία. Απαντώντας λοιπόν θα έλεγα ότι μπορείτε να βασιστείτε στην βούληση και την δέσμευσή μας. Θεωρούμε ότι έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία για την σωστή αντιμετώπιση του θέματος. Γίνεται πολλή δουλειά αυτή τη στιγμή και θα συνεχιστεί βέβαια και θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Γιάκοψαν και πάλι έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση. Όπως ακούσαμε, πολλά μπορεί κανείς να πει. Υπάρχουν ε, πολλές απόψεις, παρατηρήσεις ε, και γνώμες για το πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε τη σπατάλη τροφίμων. Άκουσα και ορισμένες ερωτήσεις, ε, στις οποίες μπορώ να σταθώ. Ξεκινώ από το ζήτημα των απολειών. Σε ό,τι αφορά την κοινή γεωργική πολιτική, Εμεί ε, συνιστούμε μόνο να συμπεριλάβουμε το ζήτημα αυτό στην ε, επικείμενη ε, αναθεώρηση πολιτική, για να δούμε πώ μπορούμε να συμβάλλει η κοινή γεωργική πολιτική και πώ μπορεί και ο πρωτογενή τομέα να αποφεληθεί από την μείωση των απολειών και τη πατάλη. Είναι σημαντικό να συμπεριλάβουμε κάτι τέτοιο στην αναθεώρηση αυτή ούτως ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι να γνωρίζουν ότι πολλοί τομείς πολιτική μπορούν να συμβάλλουν σε αυτό το εγχείρημα. Ένα άλλο ερώτημα αφορούσε την αξιολόγηση δικτύπου. Είδαμε στον ότι πώς ε, τα προγράμματα και η χρηματοδότηση ανάπτυξης της υπαίθρου μπορούν ε, να βοηθήσουν τους γεωργούς και να αυξήσουν την κερδοφορία τους. Επομένω, θέλουμε να δούμε πώς μπορούμε να περιορίσουμε τις απώλειες και ε, τη σπατάλη και πώς μπορούν επιμέρους τις ευρωπαϊκές πολιτικές να ευθυγραμμιστούν. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εξετάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την εξολόγηση του τύπου που διενεργεί, για να δει πώς μπορούν δηλαδή να ε, συντονίσει καλύτερα και πιο οργανωμένα διάφορους τομείς πολιτικής. Υπήρξε μεγάλη συζήτηση για τον ορισμό. Να προσθέσω κι εγώ ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ορισμός ε, της ε, σπατάλης τροφίμων, γιατί όπως γνωρίζετε Υπάρχει και δέσμευση έναντι του ΟΗΕ και των ε, στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Ιδίως ο στόχος 12.3 ε, κάνει λόγο ε, για τον περιορισμό κατά 50% της κατακεφαλήν σπατάλης τροφίμων και του περιορισμού των απολειών τροφίμων σε όλη την αλυσίδα παραγωγής και τη ε, επιστημική αλυσίδα μέχρι το 2030. Εγώ είμαι μόνο από το ελληνικό συνέδριο, αλλά να σας ρωτήσω πώς γίνεται να το μετρήσουμε αν δεν υπάρχει ένα σημείο αναφορά, μια αφετηρία για αυτή τη μέτρηση, για να πούν όλοι, εντάξει, εμείς κάνουμε εξοικονόμηση 20, 30, 50%. Πώς γίνεται αυτό χωρίς να έχουμε σημείο αναφοράς. Είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι σημαντικό και για τα κρατημέλη αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση της συνολό Άλλο ερώτημα αφορούσε το ζήτημα της ε, σπατάλης τροφίμων και πώς μπορεί να ιερχηθεί ψηλά στις ε, προτεραιότητες. Ε, η συνεχής πίεση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προ τα κρατη είναι ένα τρόπο, αλλά πρέπει να ζητήσουμε και από τι γενικέ διευθύνσει της να συνεργάζονται μεταξύ του για να έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Ε, να ψάξουμε να βρούμε βέλτιστες πρακτικές και παραδείγματα στα κρατημέλη. Υπάρχουν ε, πολλές ε, πρωτοβουλίες με τράπεζες τροφίμων, φιλανθρωπικά ιδρύματα κτλ. Όλα αυτά μας βοηθούν Επίσης, να αξιοποιήσουμε τις υφιστάμενες ε, δυνατότητες που μας παρέχει η κείμενη νομοθεσία. Δεν χρειαζόμαστε περισσότερη νομοθεσία, απλώς χρειαζόμαστε καλύτερη υλοποίησή της. Για να δούμε λοιπόν τι καλύτερες δυνατότητες υπάρχουν ε, στο μέλλον για να καταπολεμήσουμε τη σπατάλη. Για τις ε, δωρεές τροφίμων, με ρωτήσατε ποιοι είναι οι νομικοί περιορισμοί. Εμείς έχουμε εντάξει ορισμένα παραδείγματα στην έκθεση. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τον ΦΠΑ στα τρόφιμα. Τα κράτη-μέλη συστηματικά ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευκρινίσει πώς θα πρέπει να εφαρμόζεται ο ΦΠΑ για την χορηγία, για τις δωρεέ τροφίμων. Νομίζω ότι και αυτό θα πρέπει ε, να λυθεί επιβάλλεται φόρος προστιθέμενης αξίας ή υπάρχει απαλλαγή και πάλι όμως ε, αυτό συμμορφούται με την οδηγία ΦΠΑ. Μετά, η νομοθεσία υγειονομικού ενδιαφέροντος. Νομίζω ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένος ορισμός για το κατά πόσο οι τράπεζε τροφίμων, για παράδειγμα, θεωρούνται εμπορευόμενοι σε τον κλάδο του επιστημισμού, τότε θα πρέπει να συμμορφούνται με του ε, υγειονομικού κανόνε. Αλλά τι συμβαίνει, ισχύουν για εκείνου ή απαλλάσσονται. Πρέπει να δούμε τι ε, ισχύει και πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε προκειμένου και ε, τα φιλανθρωπικά ιδρύματα και οι τράπεζες τροφίμων να λειτουργούν πιο εύκολα. Τέλος, είναι μια ειδική έκθεση ε, του ελεγκτικού συνεδρίου. Η συνήθιση διαδικασία για μας προβλέπει ότι μέσα σε 4-5 χρόνια ε, θα επανέλθουμε και θα δούμε κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει κάτι ε, με βάση τις συστάσεις που κάναμε εμείς στην έκθεσή μας. Επομένω θα υπάρξει και συνέχεια, θα δοθεί συνέχεια στη διαδικασία αυτή για να δούμε πώς έχει επιληφθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή του ζητήματος της σπατάλης, ίσως εκπονήσουμε μια νέα έκθεση ή μπορεί να τα συμπεριλάβουμε όλα αυτά σε μια άλλη έκθεση προς εσάς για να δούμε αν έχει σημειωθεί πρόοδο σε αυτόν τον σημαντικό τομέα. Ελπίζω έτσι να έχω απαντήσει σε όλες σας τις ερωτήσεις. Ε, μπορείτε και πάλι να μου επισημάνετε να έχω ξεχάσει κάτι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους. Ας ε, περάσουμε στο επόμενο σημείο της μέσας διάταξης, ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή για το Refit των Οδηγιών για τους Οικοτόπους των Πτηνών. Είναι εδώ μαζί μας ε, ο κύριος Κρέσπο, Γενικός Διευθυντής. Να του δώσουμε το λόγο απευθείας. Ε, ζητούμε συγγνώμη για την καθυστέρηση, όμως είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση και για το προηγούμενο θέμα, όπως σίγουρα θα ισχύσει και για το δικό μας θέμα τώρα εδώ. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητά μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Με χαρά μου βρίσκομαι σήμερα ενώπιόν σας έτσι ώστε να σας ενημερώσω, να σας πληροφορήσω σχετικά με το που βρισκόμαστε σε αυτό το πολύ σημαντικό ε, χαρτοφυλάκιο για τον έλεγχο καταλληλότητα στις ε, οδηγίες για του φυσικούς οικοτόπου. Το Κοινοβούλιο ήταν πάρα πολύ ε, καλό απέναντί μας, βοήθησε πάρα πολύ. Γι' αυτό λοιπόν ήρθα εδώ να σας ενημερώσω για το πού βρισκόμαστε, ποιο είναι το state of play, τα επόμενα βήματα και για να μπορέσω να απαντήσω στις ερωτήσεις σας και να συζητήσουμε ορισμένα ζητήματα τα οποία ίσως θέλετε να θίξετε. Θα σας δείξω και ορισμένες διαφάνειες έτσι ώστε να γίνει πιο εύκολη παρουσίαση, οπότε ας αρχίσουμε. Αφετηρία, λοιπόν, δεν θα εκπλήξει κανέναν, είναι το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε με τη στρατηγική και τη βιοπικιλότητα. Και εδώ ας είμαστε ξεκάθαροι. Ο στόχος της ανάσχεσης ε, απώλειας της βιοπικιλότητας μέχρι το 2020. Στόχος της... Ε, αυτός βρίσκεται σε κίνδυνο. Στην Ευρώπη υπάρχουν πολλά ενδιαιτήματα και πολλά είδη τα οποία συνεχίζουν να ε, δείχνουν αντικές τάσεις. Μόνο το 50% των οικοτόπων έχουν σχέδια διαχείρισης, τα οποία ακολουθούνται. Το, δίκτυο, το θαλάσσιο δίκτυο Natura 2000 είναι ατελές, υπάρχουν ελλείψεις στη χρηματοδότηση και υπάρχουν επίσης περιπτώσεις ε, μη ευέλικτης εφαρμογής και ε, ανεπίτρεπτων καθυστερήσεων από τις ε, εθνικές αρχές. Επίσης υπάρχει σε γνώση, σε ανασχόληση με την εφαρμογή ε, του δικτύου και με την ε, ενημέρωση σχετικά με τα δίκτυα Natura 2000. Μόνο το 11% ε, των πολιτών γνωρίζουν τι είναι αυτά τα δίκτυα Natura 2000. Και χρειάζεται λοιπόν δράση όχι μόνο μέσα σε αυτούς τους τόπους αλλά και εκτός των δικτύων Natura 2000. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα σας εκπλήξει ο τίτλος εδώ στη διαφάνεια ότι υπό τις συνθήκες αυτές ο στόχος για το 2020 κινδυνεύει. Λοιπόν, Τι γνωρίζουμε ότι μετά τη μεγαλύτερη δημοσία διαβούλευση που έχει γίνει ποτέ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχαμε ένα τεράστιο αριθμό απαντήσεων από τους πολίτες, 552.000 απαντήσεις. Επίσης, έγινε ένας ε, δελεχέστατος έλεγχος καταλληλότητας, συλλέχθηκαν πάρα πολλά στοιχεία και είχε το Σώμα των Επιτρόπων μία συζήτηση ανατολισμού σε 7 Δεκεμβρίου του 2016, έτσι ώστε να αποφασίσει τι θα γίνει. Ήταν η πρώτη φορά που ένα τέτοιο θέμα συζητήθηκε από το Σώμα των Επιτρόπων. Το συμπέρασμα λοιπόν ήταν σαφέστατο και ήταν το ίδιο με αυτά που είπαν όλοι οι υπόλοιποι φορεί. Ότι δηλαδή οι οδηγίες ε, που αφορούν στην, ε, στους φυσικούς οικοτόπους ε, δεν θα ξανανοίξουν. Οι οδηγίες αυτές είναι καλές, είναι κατάλληλες για το σκοπό που έχουν δημιουργηθεί, όμως υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην υλοποίηση και την εφαρμογή τους. Αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημα σήμερα και γι' αυτό το συζητάμε. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε ότι έχουμε πάρα πολλά μέσα ε, υπάρχουν διεθνεί συμβάσει, υπάρχει το CBD, υπάρχει οδηγία για τα πουλιά, υπάρχουν οι στόχοι της ε, βιώσιμη ανάπτυξη, τη κύκλική οικονομία, το πρασίνισμα τη κοινή γεωργική πολιτική, οδηγία ε, για τα πουλιά, για τα ενδιαιτήματα ή του φυσικού σκοτώπου. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά μέσα που έχουμε στις διαθέσεις μα και πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε έτσι ώστε να ενισχυθεί η ε, δουλειά η αποτελεσματικότητά μα και να αναστραφούν αυτέ οι πολύ δυσίωνες ε, τάσει ε, για απώλεια τη βιοπικιλότητα. Τι αποφάσισε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι δεν θα ξανανοίξει το θέμα τη εξέταση οδηγιών, αλλά θα υπάρχουν εθνικά σχέδια που θα εστιάζουν στην εφαρμογή. Οι στόχοι αυτών των ε, σχεδίων είναι να χρησιμοποιήσουν το 100% του δυναμικού ε, του πλωστασίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προστατευτούν τα οικοσυστήματα. Τα οικοσυστήματα που ε, δεν είναι μόνο ωφέλιμα για τους πολίτες, αλλά για το περιβάλλον, για την οικονομία. Και μέσω αυτού του σχεδίου δράσης θέλουμε να συνεισφέρουμε στη στρατηγική της Ένωσης για τη βιοπικιλότητα και ταυτόχρονα να βελτιωθεί η συνοχή της οδηγίας και των υπόλοιπων οδηγιών με τους ευρύτερους κοινωνιο-οικονομικούς στόχους. Όπω σα είπα, μαζί με τις άλλες πολιτικές, δηλαδή την κυκλική οικονομία, την ενεργειακή ένωση, του αναπτυξιακού στόχου τη αυτό θα συνδυαστεί με όλα αυτά για να οδηγήσει σε πιο φιλόδοξη, αποτελεσματική και καλύτερη δουλειά, για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα και να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας για τη βιοπικιλότητα. Τέσσερις είναι οι κύριοι θεματικοί άξονες, τους οποίους θα δράσουμε έτσι ώστε να προετοιμάσουμε αυτό το σχέδιο δράσης. Οι οποίοι άξονες θα ασχοληθούν με, τα, με τις τέσσερις βασικές προκλήσεις. Καταρχάς, πρώτον, ενίσχυση της συμμόρφωσης και αύξηση της ε, πολιτικής ευθύνης. Δεύτερον, καλύτερη καθοδήγηση και ε, συνοχή με τους κοινωνιοοικονομικούς στόχους. Τρίτον, ε, υπάρχει πρόβλημα χρηματοδότηση. Δεν υπάρχουν αρκετά κονδύλια και χρειάζεται επένδυση στα δίκτυα Natura 2000 και βελτίωση των ε, συνεργειών με τα χρηματοδοτικά μέσα τη Ένωση. Και τέταρτον, χρειάζεται να γίνει τεράστια προσπάθεια σε θέματα επικοινωνία και ευαισθητοποίηση του κοινού και των ε, φορέων. Τώρα, εδώ αναφερόμαστε μόνο σε δράσεις που πρέπει να αναλυφθούν από εμάς τα επόμενα δύο χρόνια και φυσικά αυτό δεν ε, προδικάζει την ε, συζήτηση για το μέλλον της κοινή γεωργικής πολιτικής ε, και του επόμενου δημοσιονομικού πλαισίου. Εδώ δηλαδή εστιάζουμε στο ποιε είναι οι συγκεκριμένες δράσεις που μπορούμε να υλοποιήσουμε έτσι ώστε να βελτιωθεί η εφαρμογή των δύο αυτών οδηγιών. Και εδώ, στα πλαίσια αυτά, θα σας ε, ενημερώσω για κάποιες από τις δράσεις που έχουμε σκεφτεί. Καταρχάς, ενίσχυση της συμμόρφωσης και της πολιτικής ευθύνης. Ή, κάτω από αυτόν τον άξονα υπάρχουν πολλά που χρειάζεται να γίνουν. Καταρχάς, τα κράτη-μέλη πρέπει να συμπληρώσουν πλήρως και να ολοκληρώσουν τα δίκτυα Natura 2000. Αυτό πρέπει να έχει ήδη τελειώσει. Υπάρχουν ακόμα λοιπόν πολλά κενά, ιδιαίτερα ε, στη θάλασσα. Μετά, από τους 20.000 ε, οικοτόπους Natura 2000, περίπου το 80 που καλύπτουν περίπου το 80% της επιφάνειας της Ευρωπαϊκής επικράτειας της Ένωσης, μόνο το 20% από αυτά έχουν κάποια ε, κατάλληλα σχέδια διαχείρισης αυτών των ε, οικοτόπων. Εδώ υπάρχει το πρόβλημα. Ακόμα και αν όμως υπάρχει ένα σχέδιο διαχείρισης, δεν εφαρμόζεται σωστά. Μετά, χρειάζεται να γίνουν περισσότερα για την ενίσχυση της συμμόρφωσης, της ε, προώθησης ενημέρωσης και των ε, διασφαλίσεων. Όπως σας είπα υπάρχει η έκθεση ε, περιβαλλοντικής ε, υλοποίησης και εδώ θέλω να ευχαριστήσω παράλληλα και, την, ε, και εσάς, ε, την Επιτροπή Περιβάλλοντος και το Κοινοβούλιο για την προθυμία που έχετε δείξει στο να στηρίξετε αυτό το θέμα. Μετά, στα πλαίσια λοιπόν αυτού του EIR πρέπει να αρχίσουμε την, να εντείνουμε τη συνεργασία με τις άλλες χώρες για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών που θα ενισχύσουν το πλαίσιο ε, αυτό και τα δίκτυα Natura 2000. Είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε και να αναπτύξουμε περαιτέρω τα σχέδια δράσης για τα ενδυμεπτήματα και να ενισχύσουμε επίσης και τα φόρα ανταλλαγής απόψεων ε, των ε, ενδιαφερομένων. Είναι πολύ επίσης σημαντικό να υπάρχει καλύτερος διάλογος, ιδιαίτερα σε ενδιαιτήματα που, έχουν, που φιλοξενούν ταυτόχρονα πολλά ε, είδη άγρια ζωής και πανίδας, ας πούμε σαρκοφάγα, φυτοφάγα κτλ. Μετά, να σας ενημερώσω πως αυτή τη στιγμή εξετάζουμε ε, ένα πλαίσιο το οποίο αφορά τους επικονιαστές, τα έντομα αυτά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πιστεύω. Υπάρχει και, μια, και ένα συνέδριο που θα γίνει στο Κανκούν του Μεξικό, το οποίο νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό για την περαιτέρω εξέλιξη αυτής ε, της ε, πολιτικής. Οι επικονιαστές αυτή τη στιγμή είναι ένα θέμα που εξετάζουμε και προσπαθούμε να καταρτήσουμε μια στρατηγική προσέγγιση για ένα τόσο σημαντικό πρόβλημα. Όπως ξέρετε, μειώνεται δραματικά ο αριθμός των ε, επικονιαστών. Μετά, δεύτερον, χρειάζεται καλύτερη καθοδήγηση έτσι ώστε να ε, στεφθεί με επιτυχία η εφαρμογή της νομοθεσίας. Εδώ, όπως σας είπα, χρειάζεται να βελτιωθεί αυτός ο τομέας και να αφήσουμε κατά μέρους ορισμένες ε, ευφυείς ε, ας πούμε δράσεις που συνδέουν το περιβάλλον με την βιώσιμη ανάπτυξη κτλ. Αλλά χρειάζεται και επικαιροποίηση των ε, σχετικών κοινοτικών εγγράφων, διότι παρατηρούμε μια σύγχυση στα κράτη-μέλη. Δεν ξέρουν τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται, τι γίνεται, τι μπορεί κανείς να κάνει στα μέρη Natura 2000, τι δεν μπορεί. Χρειάζεται λοιπόν μια καλύτερη καθοδήγηση. Υπάρχει ανάγκη επιτακτική γι' αυτό. Και να σας ενημερώσω επίσης ότι αυτή η καθοδήγηση θα βρίσκεται στο διαδίκτυο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάνω από 20 σχετικά έγγραφα είναι ήδη διαθέσιμα και εμείς φροντίζουμε να είναι προσβάσιμα, αλλά θα υπάρχουν και ορισμένα συγκεκριμένα έγγραφα που θα αφορούν ε, πολύ σημαντικά θέματα. Επίσης, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε περισσότερους υποστηρικτικούς μηχανισμούς, κατάρτιση στις αρμόδιες αρχές, ε, ενημέρωση για τις άδειες κτλ. Η δική μου εμπειρία έδειξε από τις πολλές χώρες που πήγα ότι υπάρχει έλλειψη γνώσεων δεν είναι ενημερωμένοι για το τι περιλαμβάνει μια οδηγία, πώς πρέπει να χειριστούν την νομοθεσία κτλ. Γι' αυτό προσπαθούμε να καταρτήσουμε ε, τις αρμόδιες αρχές. Τώρα, η τεχνολογία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Ο Κοπέρνικος, οι δορυφόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούν να μας παρέχουν πολύ σημαντικές πληροφορίες για το τι γίνεται ε, στη Γη. Και μάλιστα πρόσφατα εκτοξεύσαμε δύο ακόμα δορυφόρους στα πλαίσια του Κοπέρνικος. Έτσι λοιπόν πιστεύουμε πως θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί στη διαχείριση αυτών των εκατόπων που ανήκουν στο δίκτυο Natura 2000. Τέλος, είναι πολύ σημαντικό να συμπεριληφθεί αξία των υπηρεσιών οικοσυστημάτων στον, ε, στη διαδικασία λήψη αποφάσεων και στον ε, νομοθετικό σχεδιασμό. Αυτό είναι κάτι που εξετάζουμε αυτή τη στιγμή και ελπίζουμε να το συμπεριλάβουμε στο σχέδιο δράσης μας. Τρίτος άξονας τρίτη δεσμή μέτρων είναι η ενίσχυση των επενδύσεων. Εντάξει, υπάρχει κατάρτιση, υπάρχει διαχείριση, πολύ ωραία όλα αυτά. Όμως, εάν δεν καταφέρουμε να χειριστούμε σωστά το θέμα της χρηματοδότησης, τίποτα από αυτά δεν θα πιάσει τόπο. Υπάρχει αρκετή χρηματοδότηση υπό διαφορετικά προγράμματα, είτε αυτά είναι στα πλαίσια της περιφερειακής ανάπτυξης, είτε στην αλία, την ανάπτυξη της υπαίθρου. Νομίζω κιόλα ότι μπορούμε να καταφέρουμε πολλά εάν βρούμε αυτές τις συνέργειες σε αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα και με τον τρόπο αυτό θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα προς το στόχο της βιοπικιλότητας. Επίσης, προτείνουμε τη δημιουργία αξιόπιστων δικτών που θα παρακολουθούν τις δαπάνες σχετικά με, την, ε, με τους φυσικούς ε, οικοτόπους. Πρέπει να βρούμε ένα σωστό τρόπο μέτρησης και παρακολούθησης. Και επίσης χρειάζονται μηχανισμοί που θα στηρίζουν τη χρηματοδότηση για τα δίκτυα Natura 2000 από τον ιδιωτικό τομέα. Υπάρχουν τώρα κάποιες ιδιωτικές πρωτοβουλίες, δηλαδή η χρηματοδοτική διευκόλυνση για το φυσικό κεφάλαιο, η διάφορα προγράμματα για την ε, ιδιοκτησία γης κτλ. Μετά, χρειάζεται επίσης και ε, η προώθηση στρατηγικών επενδύσεων για την αποκατάσταση της φύσης και στα πλαίσια των πράσινων υποδομών. Αυτή τη στιγμή είναι υπό εξέταση το θέμα αυτό. Υπάρχει, υπάρχει το θέμα των ε, πράσινων διαδρόμων που συζητάμε το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε με καλά αποτελέσματα θεωρώ. Και τέλος, αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να αυξήσουμε τα κονδύλια του προγράμματος LIFE. Όπως ξέρετε το πρόγραμμα αυτό έχει τρία, ε, είναι χωρισμένο σε τρία μπλοκ, την φύση, το κλίμα, το περιβάλλον. Σκοπεύουμε λοιπόν στα πλαίσια του φυστάμενου προγράμματος να αυξήσουμε κατά 10% τη χρηματοδότηση του προγράμματος που αφορά τη φύση έτσι ώστε να μην αφορά μόνο την ε, γεωργία το live, αλλά να βοηθήσει και το περιβάλλον. Προσπαθούμε λοιπόν να εντοπίσουμε πώς μπορούμε να ε, διαθέσουμε, να ανακατανύμουμε τους ε, αναγκαίους πόρους. Και τελευταίο άξονα, τελευταίο μπλοκ είναι επικοινωνία και ενδιαφέρομενοι φορεί. Όπως σας είπα, ελάχιστοι πολίτες γνωρίζουν τι είναι το δίκτυο Natura 2000. Το 95% των πολιτών είναι υπέρ της περιβαλλοντικής πολιτικής, ε, από αυτούς οι περισσότεροι πάλι θέλουν να γίνουν πολλά, αλλά μόνο το 11% από τους πολίτες ξέρει τι είναι αυτά τα δίκτυα. Και σήμερα είναι η επέτειος των, ε, της δημιουργίας των ε, δίκτυων Natura και του προγράμματος Life ταυτόχρονα, 21 Μαΐου. Και θα θέλαμε με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να δημοσιεύσουμε μία απόφαση για την θέσπιση ε, μέρας αφιερωμένης στη, στο, στα δίκτυα Natura 2000, έτσι ώστε να δώσουμε ένα μήνυμα πως είμαστε υπέρ της βιοπικιλότητας, υπέρ της φύσης, να διοργανώσουμε αρκετές εκδηλώσεις, έτσι ώστε να αυξηθεί η ενημέρωση και να δούμε πώς, ε, τι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο, πώς μπορούμε να αυξήσουμε τον ενδιαφέρον. Βλέπουμε ήδη ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τους νέους ανθρώπους. Μετά, υπάρχουν και τα βραβεία Natura 2000 που απονέμονται στις ευέλτιστες πρακτικές και στα, στην υποδειγματική διαχείριση αυτών των ε, δικτύων. Υπάρχει εντωμεταξύ τεράστια ε, ενασχόληση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό το θέμα. Τέλος. Υπάρχει μια άμεση σύνδεση φύσης και πολιτισμού. Προσπαθούμε να ε, εντείνουμε ε, και να αυξήσουμε την ενημέρωση για το πώς συνδέεται η φύση με την πολιτισμική κληρονομιά. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απεφάνθηκε ότι η Επιτροπή των Περιφερειών ε, θα μπορούσε να είναι πιο κοντά σε αυτό και να αναλάβει το θέμα ακριβώς γιατί είναι πιο κοντά στους πολίτες της περιφέρειας και να δώσει έτσι, ε, να παίξει ρόλο καθοδηγητή η Επιτροπή των Περιφερειών σε αυτές τις προσπάθειες. Τέλος, υπάρχει και το Σώμα Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, υποστηριζόμενο από το πρόγραμμα LIFE, το οποίο στόχο έχει να ε, βοηθήσει τους νέους ε, ανθρώπους που θέλουν να δράσουν εθελοντικά ή να βρουν ε, απασχόληση σε χώρο που σχετίζεται με τη φύση, με το περιβάλλον. Προσπαθούμε λοιπόν να τους βοηθήσουμε. Τίποτα όμως από όλα αυτά δεν θα γίνει αν δεν έχουμε τη δική σας βοήθεια, τη δική σας συνεισφορά. Είστε απαραίτητοι δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει, αλλά στην παρουσίαση που έκανα, τα μέτρα που ανέφερα και αυτά τα τέσσερα μεγάλα μπλοκ βρίσκονται τα περισσότερα ήδη στο σχετικό ψήφισμα του Κοινοβουλίου από το 2016. Δηλαδή, αυτό που εσείς κάνετε μας εμπνέει, αλλά επίσης αναρωτιέμαι αν έχετε και άλλες ιδέες και άλλες προτάσεις που θα μας βοηθήσουν στο έργο μας, στην κοινή μας προσπάθεια. Ποια είναι τώρα τα επόμενα βήματα. Τελευταία διαφάνεια. Έχουμε ή θέλουμε να κάνουμε ένα εθνικό σχέδιο δράσης με συγκεκριμένε δράσεις. Όχι μόνο λόγια και γενικολογίες, αλλά δράσεις συγκεκριμένες. Ας πούμε, η βιοπικιλότητα Κινδυνεύει να είμαστε λοιπόν ακριβεί, να είμαστε συγκεκριμένοι και να είμαστε πρακτικοί. Πρέπει να θέσουμε στόχους, να ξέρουμε ποιο κάνει τι και να συμμετάσχουν οι ΟΤΑ και οι χώρε μέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και όλοι οι εμπλεκόμενοι. χρονισμό τώρα για την υιοθέτηση του σχεδίου δράση είναι μέχρι το τέλο του ερχόμενου μήνα του Απρίλη. Στι 15 του Μάη θα έχουμε την έναρξη τη ημέρα του Natura 2000 και θα θέλαμε να έχουμε βεβαίω και τη συμμετοχή τη Ευρωβουλή στην ανακτήρια διάσκεψη στι 6 Ιούνιου όπου θα παρουσιαστεί το σχέδιο δράση, θα συζητηθεί με όλους τους εμπλεκόμενους για να εφαρμοστεί. Βεβαίω, ίσως και το Κοινοβούλιο θα θέλει να διοργανώσει κάποιες ακροάσεις ή εκδηλώσεις και τώρα μετά από αυτή τη συζήτηση θα θέλαμε να περάσουμε γρήγορα στη δράση, γιατί όλοι ενσυχούν για την κλιματική αλλαγή και ακόμα δεν μπορέσαμε να κοινοποιήσουμε, να μεταδώσουμε την επιτακτική ανάγκη αντιμετώπιση τη βιοπικιλότητα τη υποχώρηση τη. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε περισσότερα και σε διεθνές επίπεδο, αλλά και εδώ στην Ευρώπη. Και γι' αυτό ακριβώ Ζητάμε την δική σας την υποστήριξη, ιδέες, συμβολή. Ιδιαίτερα τώρα που ολοκληρώνουμε το σχέδιο αυτό, ώστε να υλοποιήσουμε όλα αυτά τα μέτρα επιγόντως και να βελτιώσουμε την κατάσταση, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, εκεί πρόεδρος και, και διευθυντά για την παρουσίασή σας που ήταν πολύ θετική. Εκτιμάμε την προσέγγισή σας και την Βούλη συνεργασίας με το Κοινοβούλιο ώστε να συνειδητοποιήσουν οι πολίτες μας τη σημασία της βιοπικιλότητας. Και ευχαριστούμε για τις προτάσεις σας. Και ας ελπίσουμε ότι θα κάνουμε κάτι μαζί στα πλαίσια αυτών των δύο προγραμμάτων που έχουν μεγάλη προσταμένη αξία για την Ένωση. Ο λόγος τώρα στους συναδέλφους για σχόλια. Φλόρενς πρώτα. Είστε πρώτος στον κατάλογο και στην καρδιά μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, είμαι ευγνώμων που ήρθατε, Γενική Διευθυντά, γιατί είναι πολύ σημαντικό που ήρθατε. Μα είπατε βέβαια πω ε, δεν πρόκειται να ξανανοίξουμε το θέμα τη οδηγία, ε, αλλά πρέπει να βελτιωθούν τα πράγματα. Αυτό όμω που διαπιστώνουμε δυστυχώ εδώ είναι ότι ο χώρο θέλει ζευγάρι. Και μόνο με συνεργασία μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Αλλά δεν είμαστε μόνο εμείς ε, οι εταιροί που αναφέρετε. Υπάρχουν και αγρότες, ξέρετε. Είναι και αυτοί στο παιχνίδι. Και πολλές φορές αναρωτιέμαι ε, τι μπορούν να κάνουν εκείνοι. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας ε, παροτρύνω να μην ξεχνάτε τους ε, αγρότες, τους γεωκτήμονες, όσους κατέχουν γη. Πρέπει να υπάρχει, για παράδειγμα, νομοθεσία σχετικά με την ελάχιστη απόσταση. Σε κάποιες χώρες η ελάχιστη απόσταση είναι 70 μέτρα. Υπάρχουν και άλλοι έτσι, έξυπνοι που, που έχουν θέσει τα όρια της ελάχιστης απόστασης στα 1000 μέτρα των δικτύων ε, αυτών από τις ε, κατοικημένες περιοχές και υπάρχουν βέβαια και άλλοι που δεν ε, κάνουν τίποτα απολύτω. Ε, χρειάζεται λοιπόν να δούμε τους κανόνες και να, και να φροντίσουμε έτσι ώστε να είναι συγκρίσιμοι, να μην υπάρχουν τεράστιες διαφορές. Ας δούμε για παράδειγμα τι γίνεται με το κυνήγι στην Ολλανδία. Στην Ολλανδία είναι σχεδόν απαγορευμένο το κυνήγι. Και όποιος θέλει ας πούμε, να κυνηγήσει χήνες, περιμένει στην άλλη πλευρά των συνόρων μέχρι να έρθουν οι χήνες και να περάσουν τα σύνορα και ρίχνει όσο θέλει. Γι' αυτό και σας το λέω, το έχω δει με τα μάτια μου. Και οι χήνες εντάξει, όπου προσγειώνονται ρημάζουν τα πάντα και στις περιοχές που επιτρέπεται το κυνήγι μια χαρά περνάνε οι κυπουροί και οι αγρότες, αλλά οι Ολλανδοί αγρότες οι καημένοι τραβάνε τα μαλλιά τους, δεν μένει τίποτα όρθιο. Πρέπει λοιπόν να υπάρχουν συγκρίσιμοι κανόνε, διότι δεν μπορούμε χωρί συγκρίσιμου κανόνε να πηγαίνουμε στου αγρότε μα και να του λέμε θα κάνει αυτό, θα κάνει εκείνο. Θα έχουμε πρόβλημα. Αλλά ένα πράγμα με εξοργίζει και αυτό είναι ο αγαπητός μας λύκος. Και ξέρετε γιατί, γιατί ο λύκος πάξε, μια χαρά είναι, απειλούμενο κτλ. Αλλά η Κομισιόν μας δημιουργεί προβλήματα. Υπάρχουν προβλήματα γιατί λέει ας πούμε ότι ο πληθυσμός των λύκων είναι, ε, μειώνεται, είναι είδος εξαφάνιση, πρέπει να... Ε, αλλάξει η νομοθεσία, να προστατευτεί το είδος. Στη Σουηδία όμως έχουν προσπαθήσει με πολλά προγράμματα να ε, διαχειριστούν τους επιληθισμούς και ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει απαντήσει τρεις φορές ε, στην κυβέρνηση της Σουηδίας πολύ άσχημα σχετικά με το κυνήγι των λύκων και εγώ ίδιος είμαι κυνηγός και βλέπω το πρόβλημα με τα ίδια μου τα μάτια. Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δίνει εντολές και διαταγές για το τι πρέπει να κάνει κάθε χώρα με τα ζώα της, με τους λύκους, τότε ε, στην ουσία τι κάνει, μας κάνει ε, μικροδιαχείριση, μας λέει τι θα κάνουμε στο ίδιο μας το σπίτι. Γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλώ να αφήσουμε ε, τα πράγματα που μας αφορούν σε εμά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πρέπει να εφαρμόσουμε το δίλεπτο, γιατί έχουμε πολλούς ομιλητές. Έχει κλείσει ο κατάλογος, αλλά πείτε μου. Κερπράντι, Μίλλερ και έλεγα επίσης. Ωραία, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε θα μπορούσα να συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε ο συνάδελφος Φλόρεντς. Καταρχάς, χαίρομαι για το γεγονό ότι η Κομισιόν μας εξήγησε τις προθέσεις της στα πλαίσια του σχεδίου δράσης. Εγώ είμαι μεταξύ αυτών που θεώρησαν ότι δεν χρειάζεται να ξαναρχίσουμε τη συζήτηση για όλο το πακέτο. Αυτό που χρειάζεται είναι οι μεγάλες κατευθυντήριες γραμμές να τροποποιηθούν. Και γι' αυτό το λόγο έχω μία συμπληρωματική ερώτηση σε σχέση με τα δύο κύρια κριτία που αναφέρατε. Δηλαδή, βελτίωση αυτών των μεγάλων κατευθυντήρων γραμμών που θα επανασυντάξετε. Πώς βλέπετε αυτή την αναδιάρθρωση, αν, ανασύνταξη αυτής της οδηγίας, πώς θα εφαρμοστεί. Από τη χώρα μου υπάρχουν πολλά ερωτήματα και απορίες για αυτό το θέμα και υπάρχουν κάποιες έτσι, βεβαιότητες σε σχέση με την εφαρμογή αυτών των καταθυντήριων γραμμών. Θα ήθελα λοιπόν μια ερώτηση, συγγνώμη μια απάντηση από αυτού, στην ερώτηση μου αυτή και επίσης να ρωτήσω πώς θα γίνει αυτή η διαδικασία, πώς θα εφαρμοστεί. Αν στις χώρες μέλη έχουμε ενδείξεις ότι κάποια είδη ζώων έχουν διάυξηση του αριθμού τους, υπάρχει δηλαδή θετική εξέλιξη, τότε τι θα κάνετε σε αυτή την περίπτωση. Πώς θα μεταφέρετε στην πράξη αυτή την αλλαγή. Η κυρία Μπριάνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Γενικό Διευθυντή για την παρουσίασή του. Και εγώ μεταξύ αυτών που αφενό ε, χαιρόμαστε για την... Ε, μάλλον θέλουμε να βελτιώσουμε την εφαρμογή αυτών των ε, κατευθύνων γραμμών χωρί να ξαναρχίσουμε τη συζήτηση για όλο το πακέτο. Όμω να πούμε ότι είμαστε μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση. Πιστεύω και πιστεύουμε ότι η σωστή εφαρμογή των οδηγιών, δηλαδή το γεγονό ότι κατά κάποιο τρόπο εφαρμόζεται θετικά από τις χώρες μέλη. Όλα αυτά εξαρτώ από μία λέξη, ελαστικότητα, ευελιξία. Το σχέδιο δράσης πρέπει να είναι πιο ευέλικτο σε σχέση με το παρελθόν, γιατί βεβαίως έχουν γεράσει κάποιες οδηγίες και περιβαλλοντικά τα πράγματα εξελίσσονται. Έχουμε και την αλλαγή την κλιματική, το βλέπουμε σε κάποια είδη που πριν 20 χρόνια ήταν υπερ ε, προστατευμένα, είναι ακόμα προστατευμένα ακόμα και σήμερα, αλλά ο αριθμός τους είναι αρκετά μεγάλος σήμερα, κορμοράνια ας πούμε. Εγώ ασχολούμαι και με την Αλία και ξέρω ότι αφορά και άλλους ε, συναδέλφους αυτό το θέμα και ενδιαφέρει. Ε, έχουμε τα μεγάλα σαρκοφάγα που αλλάζουν πληθυσμό του θετικά. Υπάρχουν λοιπόν ε, κάποια, άλλη, κάποια άλλα είδη, κάποια πτηνά τα οποία προστατεύονται σε κάποιες χώρες, αλλά σε άλλες χώρες όχι. Οπότε δεν γίνεται να έχουμε διαφορετική διαχείριση όπου έχουμε, σε περίπτωση όπου έχουμε ίδιες κλιματολογικές συνθήκες. Οπότε κάτι πρέπει να γίνει εδώ. Συμφωνώ να εντάξουμε και να εμπλέξουμε τους νέους, να γίνει αντιληπτό ότι είναι πολύ σημαντική η βιοπικιλότητα. Πρέπει όμως να συμμετάσχει όλος ο πληθυσμός και να μην υπάρχουν αδικίες στην εφαρμογή αυτή. Αν μετά όλα αυτά λέμε θέλουμε να τα κάνουμε, αλλά δεν διαχειριστούμε το σωστό τρόπο, απλά και μόνο οι τόποι, οι βιώτοποι η Natura 2000 ε, θα είναι κοινογράμμα. Επίσης και για την φύση υπάρχει διαφορετική ερμηνεία στις διάφορες χώρες μέλη. Κάποιες χώρες την αφήνουν ως έχει και προσεγγίζουν διαφορετικά τη Νομίζω ότι η βιοπικιλότητα έχει να κάνει με τις δικές μας ανθρώπινες δραστηριότητες, ε, τις αγροτικές, στις ορεινές περιοχές, στον νότο. Αυτή λοιπόν τη λέξη ευελιξία θα πρέπει στο σχέδιο δράση να την αναπτύξουμε από κοινού. Οπότε θα πρέπει να μου πείτε τι ακριβώ θέλετε να κάνετε σε αυτό το πλαίσιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέγει πρόεδρο. Ντόρφμαν. Σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αυτό που, τα, που είπαν οι προλαλήσαντες το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό μας είπατε πως 552.000 πολίτες συμμετείχαν σε αυτό το ερωτηματολόγιο και πως βρίσκουν την οδηγία ε, καλή κτλ. Αυτοί οι 552.000 όμως ε, δεν ξέρουμε αν έχουν επηρεαστεί από την οδηγία, μένουν ε, ή μάλλον αν έχουν επηρεαστεί θετικά. Μένουν δηλαδή σε κάποιες από τις περιοχές που ε, αφορά μέσα αυτή η οδηγία, μένουν σε αστικά κέντρα, πού ακριβώς, τι γίνεται, μένουν σε, έχουν ένα εξοχικό που πηγαίνουν κάθε εβδομάδα και βρίσκεται κοντά σε μία από αυτές τις περιοχές. Πρέπει να τα δούμε όλα αυτά για να μπορούμε να αξιολογήσουμε την αντίδρασή τους. Γιατί υπάρχουν και οι άλλοι που είναι πολύ περισσότεροι, δηλαδή που δεν έχουν απαντήσει στο ερωτηματολόγιο και ενδεχομένω έχουν τελείω διαφορετική άποψη. Σε πολλού από αυτού του ε, οικοτόπου δεν υπάρχει μόνο φύση, αλλά υπάρχουν και αγροτικέ περιοχέ, οι οποίε είναι αγροτικέ περιοχέ ε, και καλλιεργήσιμη γη εδώ και ε, αιώνε. Χρειάζεται λοιπόν να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε μια ισορροπία ανάμεσα στην ε, προστασία της φύσης και στην προστασία ε, των αγροτών. Εάν δεν υπάρχει αυτή η ισορροπία, τότε δεν πρέπει να μπορούμε γιατί υπάρχει ε, τόσο μικρή στήριξη, τόσο μικρή ενημέρωση των πολιτών για αυτή την οδηγία. Και εγώ είμαι από μια περιοχή της Ευρώπης που αυτή τη στιγμή γίνεται μεγάλη συζήτηση για αυτό το θέμα, γιατί αφορά και επηρεάζει άμεσα τους αγρότες. έρχομαι από μια, κατά κύριο λόγο, γεωργική περιοχή. Και η επέκταση του χώρου ορισμένων μεγάλων θηρευτών, όχι μόνο του Λίκου, αλλά της Αρκούδας, του Λίγκα, επηρεάσει άμεσα ε, πάρα πολλούς ε, ανθρώπους, όσους για παράδειγμα ασχολούνται με υδατοκαλλιέργειες. Γι' αυτό λοιπόν μιλάω για ισορροπία. Μην απορείτε που δεν υπάρχει θέληση των πολιτών, μην απορείτε που οι πολίτες στο δάσος όταν βλέπουν Λίκο δεν τον χαϊδεύουν ας πούμε, και δεν στέλνουν τα παιδάκια τους ε, στο σχολείο. Ε, με αυτό το, σκεπτικό. Χρειάζεται λοιπόν να δούμε το πράγμα αλλιώς. Στην Ιταλία Ιταλία, πούμε, τι γίνεται. Απόλυτη απαγόρευση του κυνηγιού λύκου, ωστόσο κάθε χρόνο ε, θανατώνονται 300 περίπου ζώα από παράνομο κυνήγι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπε και ο κύριος Φλόρενς. Χρειάζεται επικουρική αρμοδιότητα και επίσης επικουρική ευελιξία, διότι έλλειψη αυτής παρατηρούμε την ένταση και τη μεγαλύτερη αντιπαράθεση ανάμεσα σε Ευρωπαϊκή Ένωση, Κομισιόν, Βρυξέλλες και πολίτες. Και σε, πολύ, σε πολλές περιοχές της Ευρώπης το δίκτυο Natura 2000 δεν έχει κερδίσει ούτε έναν φίλο. Και αυτό πρέπει να σας το πω. Ευχαριστώ. Έχουμε πολλά να πούμε όλοι, αλλά έχουμε και περιορισμό Γεια Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριο Κρέσπο για την παρουσίασή του. Το προσμέναμε αυτό το σχέδιο δράσης. Από την αρχή, στην επιστολή στον Επίτροπο, Θέλαμε να κάνουμε ένα έτσι έλεγχο της κατάστασης της οδηγίας, της υγείας της. Να δούμε κατά πόσο το πρόβλημα οφείλεται στην εφαρμογή. Να πάντων, κάλιο αργά παρά ποτέ. Μετά από διαβούλευση με 500.000 ε, συμμετέχοντες, νομίζω ότι θα έχουμε μια πιο δυνατή φωνή. Ότι δηλαδή χρειαζόμαστε την εφαρμογή αυτού του σχεδίου δράση βάσει τη αρχική οδηγία. Για το σχέδιο δράση έχω κάποιε ερωτήσεις. Καταρχάς για τη διαδικασία. Πώς προτεθεί η Κομισιόν να εκπονήσει το σχέδιο δράση. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα, το αναφέρατε, αλλά πώ θα μπορούσε να ενταχθεί εδώ η δημόσια διαβούλευση στην εκπόνηση αυτού του σχεδίου δράση. Δεύτερον, πέρα από τις κατευθυντήριε γραμμές που αναφέρατε, τι μπορεί να κάνει η Κομισιόν ώστε να οθήσει τι χώρε μέλη να κάνουν δικά του σχέδια για τους τόπους Natura 2000 και πω η Κομισιόν μπορεί ενεργά να βοηθήσει τι χώρε μέλη στα εκπόνηση και εφαρμογή αυτών των σχεδίων δράση. Μετά, να ρωτήσω για την επιθεώρηση, τους περιβάλλοντο περιβάλλοντος, σημείο κλειδί στα πλαίσια των οδηγιών για τη φύση. Τι μπορεί να κάνει η Κομισιόν για να βοηθήσει τις χώρες μέλη ώστε να να δημιουργήσουν ένα κανονικό, ένα σωστό σύστημα περιβαλλοντικού ελέγχου. Μετά και ξέρω ότι τελειώνει χρόνος, μπορούμε να αναμένουμε ένα γενικό, μια γενική αποτίμηση και αξιολόγηση της βιοπικιλότητας και της παρουσίας της όλης της ευρωπαϊκής πολιτικής και τέλος πώς μπορεί η Κομισιόν να εντάξει στον προπολογισμό της Ένωσης τη βιοπικιλότητα. και αν υπάρχουν τέλο πάντων κάποια κονδυλία τα οποία αφορούν το πολιτέ ε, πλαίσιο και έχουν να κάνουν με την βιοπικιλότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Χάζεκαμπ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην Ευρώπη μόλις 40% της αρχικής βιοπικιλότητας παραμένει, στην Ολλανδία μόνο 15% παραμένει. Η φύση λοιπόν δέχεται μεγάλες πιέσεις από πολλούς κινδύνους, από τη ρήπανση, από την ξηρασία και βεβαίως δεν μπορούμε να περιορίσουμε την προστασία του περιβάλλοντος. Χαίρομαι που ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, διατηρεί το επίπεδο φιλοδοξίας για την υφιστάμενη ε, προστασία του περιβάλλοντος και τους οικοτόπους Natura. Πολύ συχνά θυσιάζεται η προστασία ε, του περιβάλλοντος στο βωμό τη οικονομικής δραστηριότητα και ανάπτυξης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε τώρα συγκεκριμένε ε, δράσεις και ενέργειες. Και εγώ έχω συγκεκριμένο παράδειγμα στο οποίο απαιτείται ενέργεια, γιατί στην προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να μιλήσουμε και για την προστασία των ζώων και θα πρέπει η οδηγία για τα πτηνά να ε, προστατεύει ε, τα πτηνά στην Ευρώπη. Όμως αυτό δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Εκατομμύρια μεταναστευτικά ε, πουλιά πηγαίνουν στη Μάλτα και εκεί δεν υπάρχει ούτε ξεκούραση ούτε προστασία για αυτά τα πτηνά είναι τεράστιο ο χρόνος, η ενέργεια και τα χρήματα που δαπανούν τα κράτη-μέλη για την προστασία των πτηνών και αυτό ε, δεν γίνεται στη Μάλτα. Είναι απαράδεκτες οι πρακτικές που εφαρμόζονται εκεί σε ό,τι αφορά τη θύρα ορισμένων πτηνών και η Επιτροπή ζητήσει από τα κράτη-μέλη την καλύτερη υλοποίηση της εφαρμογή, και την εφαρμογική της οδηγίας, όμως ε, δεν περιμένω ότι η Μάλτα και ως Προεδρεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ηγείται αυτής της διαδικασίας, δεν είναι αξιόπιστη η στάση της, δεν παίρνει στα σοβαρά την προστασία των πτηνών. Αυτό το Σαββατοκύριακο στη Μάλτα ε, ξεκινάει η ε, περίοδος θύρας των ορτικιών. Ζητώ λοιπόν από τους συναδέλφους να με στηρίξουν στην έκκλησή μου να δοθεί ένα τέλος σε αυτό το κυνήγι. Η Μάλτα ως Προεδρεύουσα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να ηγηθεί της διαδικασίες αυτή ε, και τη υλοποίηση τη οδηγία. Γι' αυτό σας καλώ ε, να προσυπογράψετε και εσείς την επιστολή μου στον ε, Πρωθυπουργό Μουσκάτ ε, Υπουργό Μουσκάτ. θα σας την παρουσιάσω βέβαια και θα την ε, διαβιβάσω στον ίδιο την επόμενη εβδομάδα προσωπικά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μια πολύ διαφορετική εικόνα από τις κατοχώρες. Πριν στο παρελθόν έχω υπερψηφίσει ε, την νομοθεσία για την Natura 2000, ήμουνα και στο κόμμα που τη στήριξε, αλλά με πρόδωσαν ε, μετά οι υπόλοιποι και εδώ στις Βρυξέλλες, γιατί μου είπαν ότι οι γεωργοί θα παραμείνουν γεωργοί και όχι αυτό που έχει γίνει τώρα. Αυτό δεν είναι πολιτισμική κληρονομιά. Και εδώ προς τον Γενικό Διευθυντή μπορώ να τον ρωτήσω πολύ συγκεκριμένα. Πού βρήκατε αυτά τα στοιχεία, μόνο από τις, περιβαλλοντικου τους περιβαλλοντικούς οργανισμούς, πήγατε στι ενώσεις των γεωργών στην Ολλανδία. για παράδειγμα, δεν μπορεί να, να κατασκευαστεί ολόκληρο αυτοκινητόδρομος γιατί υπάρχει ένα συγκεκριμένο ζωικό είδος ε, το οποίο απλώς ε, θυρεύεται ε, στη Γερμανία, για παράδειγμα. Ε, σε άλλε περιοχές δεν υπάρχει δυνατότητα να κάνει κάποιο ένα απλό περίπατο μέσα σε ένα τέτοιο ε, βιότοπο. Γιατί υποτίθεται ότι ε, ενοχλεί τα ζώα. Ε, αλλού στην, οι ψαράδες δεν μπορούν να πάνε να ψαρέψουν, αλλά υπάρχει κανένα πρόβλημα για τους άλλους κλάδους ε, πράσινης ανάπτυξης, υποτίθεται. Υπάρχουν λοιπόν όλες αυτές οι αντιφάσεις. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει ε, μια ισορροπία στα κοινωνικά και οικονομικά και περιβαλλοντικά ζητήματα. Στη χώρα μου δεν ισχύει αυτό. Με βάση αυτά που είπε και ο κύριος ε, Λίνς, ας μείνουμε στα βασικά, στις βασικές συστάσεις και να μείνουμε έξω από ε, τις υπερβολές γιατί αυτό το θέμα θα φέρει το τέλος της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μελιό. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχά να σα ευχαριστήσω για το ότι δεν ενώσαμε τι δύο ξεχωριστέ οδηγίε σε μία, όπω ήταν αρχική πρόθεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ευτυχώ ε, αποφασίσαμε να επικεντρωθούμε στην ε, υλοποίηση βλέπουμε πως υπάρχει ένα σύστημα το οποίο πράγματι προστατεύει τη βιοπικιλότητα και αυτό πρέπει να στηρίξουμε. Το δίκτυο Natura 2000 είναι ένα πανευρωπαϊκό σύστημα που ενώνει όλα τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορθά ε, μας λέει να, τι μπορούμε να κάνουμε για να το στηρίξουμε και να το προστατεύσουμε. Και σίγουρα είναι καλύτερο η αντιμετώπιση να γίνει σε κοινοτικό επίπεδο και όχι να αφήνουμε το κράτος μέλος να χειρίζεται την κατάσταση μόνο του ξεχωριστά. Τώρα, σε ό,τι αφορά την συμπερίληψη των ε, ενδιαφερόμενων φορέων, χάρηκα πάρα πολύ που άκουσα τις προτάσεις σας, διότι ε, ξέρετε πως υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον ε, από τους πολίτες της Ευρώπης και τους ενδιαφερμούς γι' αυτό. Και πρέπει να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσει των πολιτών, στις επιθυμίες των πολιτών. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ρωτήσω την Επιτροπή ποια είναι η αντίδρασή σας ε, σε αυτό. Ευχαριστώ κύριε Σφέλνερ. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι για αυτή τη συζήτηση και για την αναθεώρηση της οδηγίας αλλά βλέπω ότι η Κομισιόν αποφάσισε να το κάνει πλήρω. Αλλά το θέμα είναι πώ εμεί αξιολογούμε την νομοθεσία μα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να το κάνει κανεί αυτό. Ένα από του κυριότερου νομίζω είναι το πώς αυτοί που χρειάζονται την νομοθεσία μας, πώς τη βλέπουν, τι άποψη έχουν και μετά να μιλάμε για δημόσιες διαβουλεύσεις που ξέρουμε πολλές από αυτές είναι σε μια εκστρατεία να δούμε τις απαντήσεις. Αν δω τη δικιά μου την εκλογική περιφέρεια, ένα από τα πιο πολύ συζητημένα θέματα είναι η οδηγία για τους βιοτόπους, αλλά ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει. Και όπως ακούσαμε και εδώ στη συζήτηση και από την Κομισιόν και θα ακούσουμε και στο μέλλον, το θέμα είναι το πώς εφαρμόζονται όλα αυτά στις χώρες μέλη. Ωραία. Αλλά αν έχουμε τόσε δυσκολίε και τόσα προβλήματα με την εφαρμογή αυτών των διδιών, ίσως τότε οι νομοθέτε θα έπρεπε να ξανασκεφτούν το πώς γράφουν την νομοθεσία. Να αφαιρθώ σε κάτι συγκεκριμένο. Στη Στοκχόλμη, α πούμε, για τον Κορμοράνο είναι το πιο κοινό πτηνό και, και το πιο προστατευμένο υπό την οδηγία για τα πτηνά. Απαγορεύεται να τα ενοχλήσει, να τι φωλιέ, να το κυνηγήσει, να σκοτώσεις κτλ. Πολλοί όμω λένε ότι εντάξει εδώ έχουμε και εξαιρεσει υπό το άρθρο 9. Αν όμω πρέπει να εφαρμόσουμε αυτές τις εξαιρεσει, αυτές τις παρεκκλήσεις, τότε οι ψηφοφόροι και πολίτε μα, αν μάθουν ότι εμείς πρέπει να εφαρμόσουμε εξαιρέσει, τότε θα πούνε ότι κάτι πάει καλά εδώ. Αυτό θα πρέπει να το σκεφτούμε λοιπόν σοβαρά στο όλο οικοδόμημα, ότι κάτι δεν πάει καλά. Υπάρχουν κατάλογοι με ζώα που αφορούν καθαρά τη φύση, η οποία εξελίσσεται. Και θα μπορούσα να πω και ακριβώς το ίδιο παράδειγμα για τους λύκους. Το πρόβλημα είναι βέβαια ότι όλες οι σουηδικέ κυβερνήσει προσπάθησαν να προσεγγίσουν την Κομισιό να το αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα, αλλά και για του ε, λύκου και για του κορμοράνου κυνηγά την Σουηδία η Κομισιόν. Αυτό θα πρέπει να το εξηγήσουμε στου ψηφοφόρου μα, Παρόλο λοιπόν που αναγνωρίζω ότι υπάρχει ένα μεγάλο θέμα τεκμηρίωση. Αν αυτό στρέψει του πολίτε εναντίον μα, τότε θα έπρεπε εμεί να ξανασκεφτούμε το πώ γράφουμε αυτή την νομοθεσία γιατί αυτή τη στιγμή μας γεννάει μπούμεραν και μας βλάπτει. Ευχαριστώ πολύ. το θέμα. Ναι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ την Κομισιόν για την παρουσίαση. Νομίζω ότι η λέξη κλειδί εδώ πραγματικά είναι επικοινωνία. Ακούγοντας εδώ τη συζήτηση και τους συναδέλφους, εμείς δείχνουμε στις βρυξές μετά στις χώρες μέλη και δεν ξέρουμε πού βρίσκεται η ισορροπία. Είναι σημαντικό λοιπόν στο σχέδιο δράση Κομισιόν να καταστήσει σαφέστερο που βρίσκονται τα προβλήματα και πώς Κομισιών να βρούμε λύσεις και κάποια ευελιξία. Να συγχαρώ και την Κομισιόν που δέχτηκαν την πρόσκλησή μου να έρθουν στην Κομισιόν και να μιλήσουμε διάφορους φορείς όλοι μαζί, να δούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε το Natura 2000 με καλύτερο τρόπο, λαμβάνοντα υπόψη όλε τι οικονομικέ και κοινωνικέ επιπτώσει. Όπω θα δείτε, όλοι στην Ολλανδία συμφωνούν ότι θα πρέπει να έχουμε κάποια ευελιξία και μπορούν να υποβάλουν και προτάσεις για σχέδια με καλύτερη έτσι, δέσμευση και καλύτερα αποτελέσματα. Δεν ναι, θα πρέπει λοιπόν να εξετάζουμε μόνο την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, αλλά και το τι είναι δυνατό στην κάθε περιοχή. Και αυτό που με ενοχλεί και δεν μου αρέσει είναι ότι πολλέ φορέ οι ΟΤΑ λένε ότι εντάξει, αυτό είναι το γραπτό κείμενο και μα δεσμεύει από τι Βρυξέλλε. Αυτό δεν ισχύει. Οπότε εμεί ω Κοινοβούλιο και η Κομισιόν θα πρέπει να καταστήσουμε σαφέ ότι υπάρχει ευελιξία για του φορεί, ώστε να συζητήσουμε όλοι μαζί γύρω από ένα τραπέζι και να βρούμε μια κοινή λύση πιο αποδεκτή από όλου. Επίση θα πρέπει να σκεφτούμε και τους στόχους, κατά πόσο είναι ρεαλιστικοί. Όχι μόνο οι στόχοι των μονομένων χωρών μελών. Θα πρέπει να δούμε κατά πόσο θέλουμε να προστατεύσουμε τη φύση ή να αποκαταστήσουμε τη φύση στην κατάσταση που ήταν πριν χίλια χρόνια. Αυτό δεν γίνεται. Οπότε εκατοντάδες εμπλεκόμενοι θα δεχτούν σοβαρέ επιπτώσει από αυτό. Αυτό είναι ρεαλιστικό στόχος. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι επιπτώσει του κάθε στόχου και αν δεν είναι ρεαλιστικός ο στόχος πια θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε και να το αλλάξουμε. Οπότε ξαναλέω το κλειδί είναι επικοινωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σέκ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση. Ε, καλωσορίζω το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επιτέλους ε, δημοσιεύσει ένα σχέδιο δράσης. Καιρός ήταν, η κατεύθυνση που ακολουθεί είναι πιστεύω για μένα πολύ σωστή και πράγματι υπάρχουν δύο τεράστιες προκλήσεις, ε, η κλιματική αλλαγή και η απώλεια της βιοπικιλότητας. Και επιτρέψτε μου να πω ότι οι επιπτώσεις και από τα δύο είναι τεράστιες και πολύ σημαντικές. Αλλά να μην ξεχάσω να αναφέρω και τις ε, συνέπειες της εντατικής γεωργίας. Χρειάζεται λοιπόν ε, να βρούμε την αφετηρία, να ξεκινήσουμε να αλλάζουμε πράγματα. Σίγουρα πρέπει να επιτευχθεί η ισορροπία ανάμεσα ε, στην προστασία της γεωργίας και στην προστασία της φύσης. Όμως να πω επίσης ότι αυτή η ισορροπία πρέπει να αλλάξει και στο κεφάλι μας. Η ισορροπία δηλαδή για, ε, ανάμεσα στον άνθρωπο, το ζώο και τη φύση. Δεν είναι καλές οι ισορροπίες. Είναι απίστευτο να ακούω ότι ο λύκος ε, είναι κίνδυνος για τα παιδιά μας. Να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Το παράνομο κυνήγι και είναι, είναι πολύ πιο επιζήμιο για τα παιδιά μας από ότι η λύκη. Οι σφαίρες που φεύγουν αδέσποτες από τους κυνηγού ε, είναι πολύ περισσότερες και έχουν πολύ πιο βλαβερές επιπτώσεις στους ανθρώπους από ότι ένας λύκος. Υπάρχει λοιπόν μια τεράστια ε, διαφορά και οι πιθανότητες να σε χτυπήσει κεραυνός είναι πολύ μεγαλύτερες από να, σε, να σου επιτεθεί λύκος. Γι' αυτό ο κύριος ε, ο συνάδελφος που μίλησε πιο πριν είπε να μας αφήσετε να ασχολούμαστε εμείς με τα πράγματα, ε, με τα δικά μας, όμως ε, εγώ θα πω να προσέξουμε να ε, μην χάσουμε το δάσος κοιτάζοντας το δέντρο, να μην χρησιμοποιούμε αυτό το κίνδυνο του 0,001% για να νομοθετούμε λάθος. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Όκεν, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και την Επιτροπή. Χαίρομαι ιδιαίτερω. που συντάσσεστε με την ε, πλειοψηφία της Επιτροπής μας, όχι όπως παρουσιάζεται σήμερα, αλλά όπως ισχύει γενικότερα σε τη φορά του περιβάλλοντος. Νομίζω ότι Χρειαζόμαστε έναν ε, καλύτερο σχεδιασμό ίσως. Πολλοί όμως στηρίζουν μια ακόμα πιο ισχυρή ε, για παράδειγμα, στην, περιφέρεια, στην Επιτροπή των Περιφερειών ήθελαν μια ακόμα ισχυρότερη εφαρμογή και υλοποίηση του Natura 2000. Επομένω, το ποιον εκπροσωπούμε και ποιος εκπροσωπεί τον λαό, δεν ξέρω. Ο καθένας εκπροσωπεί τους ψηφοφόρους του. Μόνο αυτό μπορούμε να πούμε. Στο Παρίσι συνάντησα τον Γενικό Διευθυντή της ε, Σύμβασης Βιοπικιλότητας του ΟΗΕ, τον κ. Ντίας, και ανέφερε ότι η βιοποικιλότητα είναι εξαιρετικά σημαντική και για το κλίμα. Βέβαια και το κλίμα είναι πολύ σημαντικό για τη βιοπικιλότητα, αλλά και η βιοπικιλότητα συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό ε, σε ό,τι αφορά τι εκπομπέ του διοξιδίου του άνθρακα. Και έτσι όλα αυτά βοηθούν ε, τον περιορισμό τη κλιματική αλλαγή. Είναι κάτι το οποίο δεν αναφέρεται, δεν αναφέρθηκε σχεδόν καθόλου στο Παρίσι. Όμω πρέπει και αυτό να το λάβουμε υπόψη. Η βιοπικιλότητα ωφελεί τη διάσωση του κλίματος και μετά για τη χρηματοδότηση. Εγώ ασχολούμαι με αυτό το ζήτημα εδώ για μια δεκαετία εδώ στο Κοινοβούλιο και είναι πολύ δύσκολο ε, να πείσουμε ένα κράτος μέλος ε, να δαπανίσει τα απαραίτητα κονδύλια αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει τα δέοντα. Τι μπορούμε να κάνουμε. Όλα αυτά τα χρήματα που διοχετεύουμε στην κοινή γεωργική πολιτική, να πούμε τουλάχιστον ένα τμήμα τους θα πρέπει να συνδέεται με το γενικό συμφέρον ε, με υποχρεωτικό τρόπο και όχι εθελοντικό. Αυτό αν θέλουμε να κάνουμε όσα μας αρμόζουν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκοστέτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και την Επιτροπή για τις εξηγήσεις που μας έδωσε προηγουμένως. Θεωρώ ότι αυτές οι δύο οδηγίες για τα πτηνά και τα οικοσυστήματα είναι θεμέλιος λήθος ε, της ευρωπαϊκής πολιτικής για την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας που είναι σημαντική τομή. Γι' αυτό και η εφαρμογή τους θα πρέπει να παρακολουθείται εκ του σύνεγγης, όμως ε, αυτό αυτά τα κείμενα δεν ε, τίθενται ένα αμφιβόλο. και εγώ στο παρελθόν, στην πράξη, ε, είχα τη δυνατότητα και την ευκαιρία να εφαρμόσω στην πράξη αυτές τις δύο οδηγίες και νομίζω ότι τα ωφέλη υπερβαίνουν ε, τα υπέρ και τα κατά που ε, αναφέρουμε για αυτές τις δύο οδηγίες. Όμως θεωρώ ότι η εφαρμογή των οδηγιών νομίζω ότι απαιτεί και κάποια ευελιξία για να λάβουμε υπόψη την ιδιαιτερότητα της επικράτειας. Ε, τη βούληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, να διορθώσει τις ελλείψεις και αδυναμίες ε, σε ό,τι αφορά τις δύο οδηγίες. Νομίζω ότι το σχέδιο δράσης είναι κάτι το θετικό, όμως πρέπει να μιλήσουμε και πάλι για το λύκο. Γιατί υπάρχουν ασυνέπειες ε, στο παράρτημα τη οδηγία των οικοσυστημάτων, γιατί δεν λαμβάνουμε υπόψη την περιφερειακή διάσταση του ζητήματο και η υλοποίηση των οδηγιών χωρίς καμία ευελιξία έχει οδηγήσει σε μεγάλη άνοδο ε, των, ε, των ολίκων, σε μεγάλη άνοδο του αριθμού τους, σε βάρος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και βέβαια επεκτείνονται όλα και περισσότερο και σε άλλες ε, γαλλικές ε, περιοχές και δημιουργεί τοπικές εντάσεις. Να γνωρίζουμε ότι δεν πρόκειται μόνο για θηρευτές. Δεν μπορούμε να ε, κυνηγήσουμε τον λύκο εκτός και αν υπάρχουν συγκεκριμένες άδειες. Αυτό όμως λειτουργεί αρνητικά και για τον τουρισμό. Θα ήθελα λοιπόν, στρεφόμενοι προς την Επιτροπή, να μου πείτε περισσότερα σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη αυτού του σχεδίου δράση για τι αδυναμίε που θα καλύψει και τι ελλείψει και, ελλείψεις και τι συμβαίνει πιο συγκεκριμένα στην περίπτωση του Λίκο Ευχαριστώ, ευχαριστούμε και εμεί. Ο κ. έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που βλέπω όλου αυτού του συναδέλφου να παίρνουν τον λόγο να συμμετέχουν σε αυτή τη συζήτηση για την φύση και την βιοπικιλότητα, γιατί έχει πέρασει καιρό από την τελευταία φορά που συνέβη αυτό. Η κυρία Σκράγια Πύρικ ε, με έχει απογοητεύσει, γιατί δυστυχώς ε, η Γενική Διεύθυνση τώρα δεν μπορεί να απαντήσει στις ψευδεί ε, καταγγελίε, γιατί αποχώρησε η ίδια. Πρώτα απ' όλα είναι σημαντικό να κάνουμε μια διάκριση ε, μεταξύ ορισμένων περιστατικών και της ευρύτερη εικόνας. Ε, μίλησαν λοιπόν για συγκεκριμένα περιστατικά για τους κορμοράνους, τους λύκους και το καθεξής. Υπάρχει περιθώριο ευελιξία στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και νομίζω ότι ε, πολύ σωστά αναφέρθηκε προηγουμένω ε, ότι αν κάποιο θέλει να βρει την ευελιξία σε περιφερειακό επίπεδο, τη βρίσκει και βρίσκει και λύση μεταξύ των φίλων του περιβάλλοντος, των γεωργών και το καθεξής. Όλα αυτά υπάρχουν όμως. Ας δούμε την ευρύτερη εικόνα. Το 2011 αξιολογήσαμε την προηγούμενη στρατηγική για την ε, βιοπικιλότητα και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι απέτυχε παταγωδός. Η νέα στρατηγική για την βιοπικιλότητα μέχρι το 2020 είχε τον ίδιο στόχο να ανακόψει ε, την ε, απώλεια της βιοπικιλότητας, αλλά χάρη, ανέφερε μάλλον Γενική Διεύθυνση, και να αποκαταστήσει τα οικοσυστήματα στο βαθμό του δυνατού. Δηλαδή, αν δεν, έχει, δεν έχουν υποστεί τα οικοσυστήματα αυτά, μία αναστρέψιμη ζημία. Πάμε λοιπόν ακόμα παραπέρα. Τώρα, με την ενδιάμεση αναθεώρηση, γνωρίζουμε ότι η κατάσταση είναι απελπιστική. Δεν θα τα καταφέρουμε. Είναι πρόβλημα? Βεβαίως και είναι. Γιατί η βιοπικιλότητα είναι αυτή που αποτελεί ε, θεμέλιο λίθο και της οικονομικής μας δραστηριότητα σε ό,τι αφορά το νερό, ε, το, το έδαφος, ρυθμίζει το κλίμα, μας προστατεύει από ακραίες καιρικές συνθήκες, μας επιτρέπει να ζούμε ως ε, ανθρώπινο είδος. Και αυτό, αυτά τα αντλώ από την πρώτη πρόταση της ανακοίνωσης της Επιτροπής. Αυτό είναι το διακύβευμα λοιπόν όχι συγκεκριμένα ήδη για περιστατικά, το μέλλον μα ε, ως ανθρωπότητα. Το 2011 λοιπόν υιοθετήσαμε την έκθεσή μου για την αξιολόγηση και για το μέλλον τη στρατηγική τη βιοπικιλότητα, η οποία μάλιστα υπερψηφίστηκε ομοφόνο από αυτή την Επιτροπή. Α ε, διατηρήσουμε λοιπόν, α μείνουμε σε αυτέ τι δεσμεύσει προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα, πότε να περιμένουμε το πρόγραμμα εργασιών για τη χρηματοδότηση πολύ λίγα γνωρίζουμε για τα ε, μέσα χρηματοδότησης στα κράτη-μέλη. Δώστε μας επιτέλους μια εικόνα, γιατί δεν ξέρουμε τίποτα. Και τι συμβαίνει με την γεωργική πολιτική. Ο Φιλ Χόγκαν ε, είναι πλήρως αφοσιωμένος στην βιοπικιλότητα ή όχι. Πράγματα απλούστατα, όπως η μη χρήση ζυζανιοκτώνων ε, στις χώρες, ε, συγγνώμη, περιοχές συγκεκριμένου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντο θα έπρεπε να έχει λυθεί εδώ και καιρό. Τελικά είναι θέμα επιλογών. Και αυτή την πολιτική πρέπει να κάνουμε και εμείς ως πολιτική. Είναι θέμα της ευρύτερη εικόνας λοιπόν. Ευχαριστώ. Επιλογές και κανόνες να προσθέσω εγώ. Έχουμε συμφωνήσει για δύο λεπτά μόνο. Να παρεμβαίνετε κυρία Γκέλινγκ. Ευχαριστώ. Πολλοί προηγούμενοι ομιλητές έχουν πει περίπου αυτά που ήθελα να πω κι εγώ. Μία παρατήρηση μόνο. Είναι αλήθεια ότι δεν δίνουμε αρκετή αξία στη βιοπικιλότητα. Θα δείτε ότι δεν καταβαίνουν πολλοί σε για τη βιοπικιλότητα. Κάποιοι το κάνουν, αλλά όχι αρκετοί. Και εγώ για να σας υπενθυμίσω το δίδαγμα του Brexit Μπορώ να σας πω ότι αυτό το θέμα δεν ετέθη επιτάπητος προ-Brexit. Σίγουρα όμως γίνεται τώρα όταν ε, κάποιοι θεωρούν ότι απειλείται η βιοπικιλότητα ε, και η προστασία της. Είναι το ερώτημα που μου θέτουν πιο συχνά. Αυτό εν είδη προειδοποίηση ότι θα ήταν πολύ καλό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταβάλει μεγαλύτερε προσπάθειε ε, για να ξεκαθαρίζει και να διαφημίζει ουσιαστικά το τι ε, έχουμε. Γιατί όπως λέει και η Τζονι Μίτσελ, δεν ξέρουμε τι έχουμε μέχρι να το χάσουμε. Ευχαριστώ κυρία Μιλέρ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ βλέπω με μεγάλη μου χαρά πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιμένει στο να υπάρχουν δύο ξεχωριστές οδηγίες και ε, πως μάλιστα έχει διατυπώσει συγκεκριμένες σαφείς προτάσεις. Θα ήθελα όμως ε, να ρωτήσω ποια είναι τα κρατη που δεν έχουν εφαρμόσει τις οδηγίες αυτές. Είναι γνωστό πως ορισμένα δεν είναι σε θέση ε, να το κάνουν. Μετά η ευελιξία είναι κάτι που αναφέρθηκε ήδη και οι κάτω χρησιμοποιούν τις ε, περιοχές του δικτύου Natura 2000. Ε, βλέπουμε ότι υπάρχουν θέματα με το λιμάνι του Ρότερνταμ και πρέπει να, αλλάξει, πρέπει να αλλάξουν τα όρια λόγω των ε, περιοχών Natura 2000. Όμως υπάρχουν και οι ορεινές περιοχές και εγώ προσωπικά προέρχομαι από μια τέτοια εποχή και εμείς επηρεαζόμαστε άμεσα από την οδηγία αυτή η βιοπικιλότητα έχει διατηρηθεί όλα αυτά τα χρόνια που εμείς ε, καλλιεργούμε ε, τη γη στην ε, πατρίδα μου, αλλά από την άλλη τώρα μας περιορίζει η νέα οδηγία. Υπάρχουν λοιπόν διάφορες πτυχές του ίδιου θέματος και όπως είπε και ο κύριος Γκερμπράντι δεν πρέπει να τις παραβλέπουμε. Και εμείς ε, επίσης στις ορεινές περιοχές έχουμε σοβαρά προβλήματα με τους ε, κορμοράνους, με τους κόρακες, με τις κουρούνες, με τους λύκους, ε, τα οποία ζώα αυτά όταν ζουν σε απικίες θέτουν σε κίνδυνο το βιός μας, τις καλλιεργίες μας. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται ευελιξία. Και να πω τώρα κάτι και για τους μεγάλους θηρευτές, για το λύκο κτλ. δεν είναι θέμα αν θα επιτεθεί ο λύκος σε άνθρωπο. Το θέμα είναι ότι ε, όπου ζει ο λύκος ε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε τη γη, δεν ε, μπορεί να σωθεί η βιοπικιλότητα που λέτε. Το αντίθετο εξαφανίζονται όλα τα λαζόα. Η βιοπικιλότητα, ξέρετε, δεν είναι μόνο λύκος, είναι και ένα φυτό, ένα λουλούδι. Γι' αυτό λοιπόν αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και πρέπει να ζυγίσουμε τα πράγματα και να δούμε τι είναι πιο σημαντικό. Ένα ζώο ή ε, καλλιέργεια που ε, σώζει και δίνει τροφή σε ολόκληρη κοινωνία. Ευχαριστώ κύριε Φιτικάινεν. Πρώτον, για την απώλεια τη βιοποικιλότητας είναι ακόμα μεγαλύτερη απειλή από την κλιματική αλλαγή. Πρέπει να το πάρουμε λοιπόν πολύ στα σοβαρά. Για τους λόγους που έχουμε ήδη ακούσει. Και μετά, αυτές οι δύο οδηγίες δεν πετυχαίνουν τον τελικό στόχο και χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δεσμεύεται να γίνει καλύτερο θεματοφύλακα της ε, υλοποίησει τους. Μετά, σε ό,τι αφορά την ευελιξία, ήδη υπάρχει ευελιξία, για παράδειγμα με τους Υπάρχει άδεια ε, για κάποιον να τους κυνηγήσει και να τους σκοτώσει, αν είναι απειλή για ανθρώπους ή για την οικονομία. Μετά, για υποχρεωτικές δράσεις. Όπω συμβαίνει με του φόρου. Ε, είναι υποχρεωτικό να πληρώσει φόρου, δεν χρειάζεται να του ρωτήσουμε αν του αρέσει ή όχι. Κάποιε φορέ γίνεται όμω. Και αυτό γιατί, γιατί ε, άλλοι θα αναλάβουν το κόστος αν δεν ε, ενεργήσουμε εμείς. Αυτό συμβαίνει και με την προστασία των ζώων, του περιβάλλοντος και της χλωρίδας ε, και πανίδας. Βεβαίως και πρέπει να διαφυλάξουμε ε, τον ε, κανονισμό. Στη Φιλανδία. Η πολιτική κατά, ενάντια μάλλον σε έρευνες και μελέτες, προχώρησαν σε ενέργειες για τους λύκους. Υπάρχει σοβαρό ζήτημα. Επομένω, προς την Επιτροπή μπορώ να ρωτήσω αν επιτέλους θα αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις για την υλοποίηση και να ασκήσει κυρώσεις στις ε, χώρες που δεν ε, εφαρμόζουν τις οδηγίες όπως πρέπει. Ευχαριστώ. Να δώσουμε τώρα το λόγο στον Γενικό Διευθυντή. Μεγάλο το ενδιαφέρον, αλλά νομίζω ότι λίγο υπήρξε μια επανάληψη συγκεκριμένων ε, θεματικών τομέων. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και όλα τα μέλη, γιατί από τη συζήτηση ξεκάθαρα προκύπτει ότι είναι πολύ σημαντικός ο φάκελος αυτός. Έχετε γύρει πολλά ζητήματα και δεν με εκπλήσει αυτό, γιατί εξετάζουμε κάτι το οποίο είναι θεμελιώδη σημασία. Η προστασία της βιοπικιλότητας σημαίνει και η προστασία του πλανήτη μας. Και πολλά μέλη ανέφεραν και πώς επηρεάζεται έτσι και η κλιματική αλλαγή. Ε, πρόκειται για την καθημερινή ζωή των ε, συμπολιτών μας. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε επιμέρους ζητήματα που έχετε θίξει. Κάποιο ανέφερε ποιο έχει απαντήσει, ποιον τον ενδιαφέρει αυτό το ζήτημα. Όλος μας αφορά. Δεν είναι θέμα του ενό ή του άλλου γεωργού ή κάποιε περιβαλλοντικέ οργάνωση. Όλου του πολίτε του αφορά η του αλλου γεωργου η καποιε περιβαλλοντικε οργανωσει ολου του πολιτε του αφορα η στρατηγικη για την βιοποικιλότητα. Και γι' αυτό για πρώτη φορά στην ιστορία τη Ευρωπαϊκή Ένωση είχαμε πάνω από 500.000 απαντήσει. Πολίτε που μα είπαν ότι αυτό είναι σημαντικό για μα. Εντάξει, σε πολλέ περιπτώσει ήταν ενώσει, σύλλογοι, ομοσπονδίε, αλλά πολλέ φορέ ήταν και απλοί πολίτε που μας είπαν είναι σημαντική η βιοπικιλότητα. Δεν θέλουμε να περιοριστεί ε, το επίπεδο της προστασίας, ε, ούτε να ξανανοίξει η διπραγμάτευση για, τους, ε, για τις οδηγίες, ούτε να υπονομεύσουμε το σύστημα το οποίο έχει θεσπιστεί μετά από τόσο κόπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρουμε ότι υπάρχουν προβλήματα προς, ως προς την εφαρμογή, όμως ας λύσουμε πρώτα αυτό το θέμα της εφαρμογής, ας βρούμε κάποιες καλές λύσεις για τη χρηματοδότηση, τα διαχειριστικά σχέδια. Ας συνεργαστούμε με τις περιφέρειες, τις τοπικές αρχές, αλλά σας παρακαλώ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να μην υποβιβαστεί το επίπεδο προστασίας ή η φιλοδοξία σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της απώλειας ε, βιοποικιλότητας, Γιατί σε αυτή την περίπτωση θα έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα για την ευημερία μας, για την οικονομία μας για όλους τους ε, πολύ σημαντικούς στόχους ε, που πολύ σωστά υπενθύμησε και ο κύριος Γεμπράντη. Πολλά ερωτήματα, θα προσπαθήσω να απαντήσω. Πρώτον, για τους γεωργούς. Αν έχει υπάρξει διαβούλευση με τους γεωργούς, αν έχουν συμμετάσχει, μάλιστα, είχαμε εκτενέστατες διαβουλεύσεις, μάλιστα, με τις ε, ενώσεις παραγωγών, γεωκτημόνων, και το σχέδιο δράσης ε, θα συμπεριλάβει και πλατφόρμες σε διαλόγου με τα διάφορα μέρη. Θα υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας με τις ε, τοπικές κοινότητες για ε, την διευθέτηση τέτοιων ζητημάτων. Θέλουμε να συνεργαστούμε και με τους γεωκτήμονες, ούτως ώστε η επίτευξη των στόχων να συνάδει και με την επίτευξη κοινωνικο-οικονομικών στόχων. Αυτό το αναφέρουμε και στις οδηγίες και θα διατηρήσουμε τη δέσμευσή μας ότι αφορά τις συζητήσεις ε, με όλους ε, τους ευλεκόμενους ε, κλάδους οικονομίας γιατί θέλουμε οι λύσεις που θα βρούμε να ωφελήσουν και την τοπική κοινωνία. Από πολλές παρεμβάσεις διαπίστωσα μία αντίφαση μεταξύ του Natura και τη οικονομική δραστηριότητα. Νομίζω ότι ένα από τα μηνύματα του Natura 2000 και τη βιοποικιλότητας είναι ότι η προστασία τη βιοποικιλότητας δεν είναι κάτι το ασύμβατο ε, με την οικονομική δραστηριότητα. Οικοτουρισμός. Βιώσιμες ε, αγροτικές πρακτικές. Υπάρχει τρόπος να προστατεύσουμε και το περιβάλλον, αλλά και να έχουμε οικονομική ανάπτυξη και οι βλεκόμενοι φορείς, ε, οι κατεξοχήν ενδιαφερόμενοι, είναι οι γεωργοί. Γιατί όσο λιγότερο επενδύουν στη βιωσιμότητα, τόσο υπονομεύουν ε, τα περισσότερα του στοιχεία, τόσο ε, οικονομική δραστηριότητα θα έχουν τελικά. Πρέπει να τα συζητήσουμε όλα αυτά, να δούμε ποιες λύσεις θα βρούμε. Πολλά τα, ερωτήματα για την ε, καθοδήγηση. Το ανέφερε ο κ. Λίνς, υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα. στους μισούς ε, οικοτόπους ε, του Natura 2000 δεν έχουμε κα, κανένας είδους διαχείριση. Επομένως, μπορεί να υπάρχουν παράπονα ότι δεν ε, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Ναι, αλλά άμα δεν υπάρχει διαχειριστικό σχέδιο, είναι πολύ δύσκολο να διασφαλίσει κανείς μια βιώσιμη διαχείριση. Γι' αυτό και θα εργαστούμε για να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη, τις τοπικές και περιφερειακές αρχές για να έχουν ε, σωστά διαχειριστικά σχέδια. Αυτό πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα. Δεν γίνεται μόνο 50% των ε, βιοτόπων να έχουν ε, τέτοια σχέδια και τα υπόλοιπα όχι. Θα βασιστούμε και στην υφιστάμενη καθοδήγηση και τις γραμμές. Θέλουμε όμως να τα επικαιροποιήσουμε και να τα αναβαθμίσουμε για να ανταποκριθούμε σε προβλήματα που έχουμε εντοπίσει στον έλεγχο καταλληλότητα. και ε, έχουμε την πρόταση να το κάνουμε αυτό με όλους τους εμπλεκόμενου φορείς. Γι' αυτό η Επιτροπή των Περιφερειών ε, βρίσκεται σε στενή επαφή μαζί μα και έχουμε και τους ε, αρμόδιους επιτρόπους αλλά και εκπροσώπους από την Επιτροπή των Περιφερειών. Και εγώ μάλιστα έχω πάει στην Επιτροπή των Περιφερειών να τους παρουσιάσω τις πρωτοβουλίες και να ζητήσω την ε, συμμετοχή τους στο τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Κάποια από τα μέλη της Επιτροπής επίσης αναφέρθηκαν στην ευελιξία. Κάποιοι λένε ότι είναι πολύ αυστηρή η νομοθεσία και άκαμπτη και ότι ίσως ε, πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερο περιθώριο ευελιξίας και ελαστικότητας. Εγώ θεωρώ ότι το σχέδιο δράσης θα δώσει αυτή την ευελιξία, πάντα με σεβασμό προς τους κανόνες και αυτή η ευελιξία μπορεί να επιτευχθεί δίνοντας καθοδήγηση σε ό,τι αφορά την ερμηνεία των νομικών διατάξεων. Όμως όταν αποφασίσουμε ότι δεν θα ξανανοίξουν ε, οι οδηγίες, δεν γίνεται κάτι άλλο. Μπορούμε απλώς να τις εξετάσουμε, να τις συζητήσουμε τι συμβαίνει στις επιμέρους επικράτειες, περιφέρειες, τοπικές κοινωνίες, αλλά πάντα ε, με σεβασμό προς ε, το νομικό καθεστώς. Ο κύριος Ντόρφμαν τώρα ρώτησε για τα διαχειριστικά σχέδια, πώς οι πολίτες ε, εμπλέκονται, απάντησα. Ο κύριος Γιαβόρ ζήτησε περισσότερες πληροφορίες στη διαδικασία. Για το χρονοδιάγραμμα πρώτα απ' όλα, είπα αν όλα πάνε καλά, το σχέδιο θα είναι έτοιμο μέχρι τα τέλη Απριλίου. Τον επόμενο μήνα λοιπόν. Η δημόσια διαβούλευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Και τώρα βάσει του ε, σχέδιου δράσης ε, θα εξετάσουμε τι καθοδήγηση έχουμε, πού πρέπει να επικαιροποιηθεί και πού χρειάζονται περισσότερες ε, οδηγίες πάντα κατόπιν διαβούλευσης και ε, με τα Τώρα, επιθεωρήσεις και επιβολή της νομοθεσίας. Η κυρία είναι αναφέρθηκε σε αυτό. Έχουμε την πρωτοβουλία για την διασφάλιση της συμμόρφωσης. Ε, στο EIR έχουμε εντοπίσει ε, το Nature ως συγκεκριμένο κλάδο. Θα συνδράμουμε τα μέλη που υπάρχουν προβλήματα και αν σε ορισμένε περιπτώσει υπάρχουν παραβιάσεις ε, της νομοθεσίας... θα προχωρήσουμε βεβαίως. Γιατί πρέπει να γίνονται σεβαστές οι οδηγίες, παρότι δεν θα ξανανοίξει η εξέτασή τους. Όταν υπάρχει λοιπόν ε, παράβαση, κινούμε τις απαραίτητες διαδικασίες. Επειδή είμαστε θεματοφύλακες ε, των συνθηκών σε αυτό το τομέα, ο κύριος Γιαβόρ, μήπως θα μπορούσαμε να εντάξουμε τη βιοπικιλότητα σε κάθε τομέα 20% του προπολογισμού αφορούν στην κλιματική αλλαγή. Τίποτα αντίστοιχο όμω δεν ισχύει για τη βιοπικιλότητα. Πώ θα μπορούσε αυτό να γίνει στο επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Το είπα και στην αρχή τη παρουσίασή μου, ότι εμεί δεν προκαταβάλουμε δεν προδικάζουμε το επόμενο πι δελτα πι, όμως υπάρχουν πολλά που μπορούν να επιτευχθούν με ε, τους υφιστάμενους πόρους, με το life, αυξάνοντας το ποσοστό του nature ε, και με τα διάφορα ταμεία. Αν μετά το 2020 υπάρχει πολιτική συμφωνία για να δοθούν συγκεκριμένα κονδύλια στη βιοπικλότητα, αυτό θα ήταν ε, πολύ καλά νέα. Όμως εμείς επεξεργαζόμαστε αυτό το σχέδιο δράσης για να έχουμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες τα επόμενα χρόνια, χωρίς να προδικάζουμε το μέλλον του ΠΔΠ. Μετά, ερωτήσεις για συγκεκριμένα είδη, ε, πτηνά, κορμοράνι, λύκη και τι κάνουμε. Εδώ θα ήθελα να πω ότι η οδηγία για τα πτηνά ήδη παρέχει περιθώριο ευελιξίας ε, για να αντιμετωπίσουμε διάφορα τέτοια προβλήματα. Η Επιτροπή έχει δώσει οδηγίε σε πολλού τομεί και καθοδήγηση. Όμω θα πρέπει και τα κράτη-μέλη να αναλάβουν τι ευθύνε του. Όταν υπάρχει ένα δύσκολο πρόβλημα με την τοπική κοινωνία, κάποια στιγμή, κάποιε φορέ μάλλον, αντί να αξιοποιούν την ευελιξία που του παρέχεται για να αντιμετωπίσουν το ζήτημα, ε, βλέπουμε ότι το αρίχνουν όλα στι Βρυξέλλες. ρίχνουν το φταίξιμο λοιπόν στις Βρυξέλλες και νομίζω ότι πρέπει να γίνει καλύτερη δουλειά με τις τοπικές κοινωνίες ε, για τη λύση των ε, προβλημάτων. Δεν θεωρούμε ότι το πρόβλημα είναι η έλλειψη ευελιξίας των οδηγιών. Υπάρχει έλλειψη διαλόγου κάποιες φορές, ε, ελληματική ή ελλειπής μάλλον εφαρμογή και υλοποίηση και συμβατότητα μεταξύ της επιβολής του νόμου και της προστασίας να λάβουμε υπόψη βέβαια και τυχόν ε, προβλήματα, όμως οι οδηγίες επιτρέπουν ε, στα κρατημέλη να αναλαμβάνουν τις απαραίτητες ε, ενέργειες όταν υπάρχει σοβαρή ζημία ως προς το περιβάλλον ή ως προς το προστατευόμενο είδος ή ως προς την τοπική κοινωνία. Επομένω, υπάρχει στην ουσία των οδηγιών αυτών αυτή η φιλοσοφία συμφιλίωση των δύο ζητημάτων. Εμείς ε, σε ό,τι αφορά την πιο περιοριστική υλοποίηση των οδηγιών, όχι δεν το επιθυμούμε. Εμεί θέλουμε πιο αποτελεσματικά να υλοποιείται το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και να υπάρξει ισορροπία μεταξύ της ασφάλειας δικαίου, της δικαιοσύνης και της ευελιξίας. Κάποιοι ευρωβουλευτέ ε, ρώτησαν ε, τι συμβαίνει με τι ιδιομορφίε του κάθε κράτου μέλου. Βεβαίω, αν το σχέδιο δράση υλοποιείται. Αυτό πρέπει να γίνει μόνο με σεβασμό προς τις ιδιομορφίες του κάθε κράτους μέλους και έτσι εδώ εκτιμούμε ιδιαίτερως και τη στενή συνεργασία με την Επιτροπή των Περιφερειών και έχουμε και την πρόθεση να λάβουμε υπόψη ε, όλες ε, τις κοινωνικές, οικονομικές ε, και πολιτισμικές περιποθέσεις καθώς και τα τοπικά χαρακτηριστικά κάθε επικράτειας. Οι διμερεί διάλογοι που θα διοργανώσουμε με τα κράτη-μέλη θα μα βοηθούσαν με καλύτερο τρόπο να εκτιμήσουμε τι ανάγκε και να βρούμε ε, τις λύσεις που επιθυμούμε. Τώρα, κάποιες ε, ερωτήσεις αφορούσαν τη διεύρυνση του Natura 2000. Τι συμβαίνει με τα μεταναστευτικά είδη, όταν ξεπερνούν δηλαδή την οριοθέτηση. Νομίζω ότι η βασική ιδέα του Natura 2000 αφορούσε τη δημιουργία ενός δικτύου, ενός δικτύου προστασίας της βιοποικιλότητας. Και νομίζω ότι και η έννοια της βιογεωγραφίας, ε, των υπηρεσιών οικοσυστημάτων, των πράσινων υποδομών θα ενταχθούν στο σχέδιο δράσης για να διευκολύνουν ακριβώς αυτή την προσέγγιση δικτύου. Ο κύριος Χέτεμα μίλησε με ιδιαίτερη έμφαση για την ε, σημασία της επικοινωνίας. Και εδώ και εγώ πιστεύω ότι είναι από τους ε, βασικούς άξονες. Επικοινωνία με τους ε, πολίτες, με τους εμπλεκόμενους φορείς, με τις τοπικές αρχές. Για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, τα περισσότερα ήδη αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη βρίσκονται σε φθήνουσα πορεία ε, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα, αλλά αυτό να γίνει πάντα σε συμφωνία με τις τοπικές κοινωνίες, με ε, τους εμπλεκόμενους φορείς, τις περιφέρειες και τα κρατημέλη. Υπάρχουν και δύσκολα ζητήματα και περιπτώσεις και εμείς ε, δεν θα το αποφύγουμε. Και εγώ προσωπικά έχω πάει σε πολλούς ε, χώρους ε, του Natura 2000, έχω μιλήσει, συνομιλήσει με τις τοπικές αρχές για τα προβλήματα αυτά και για τις λύσεις. Υπάρχουν και λύσεις που συμμορφούνται πλήρως με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, όμως θα πρέπει να υπάρχει και η βούληση εξέβρεση των καλύτερων λύσεων, της χρηματοδότησης που απαιτείται και ούτω καθεξής, λαμβάνοντας υπόψη και τα συμφέροντα και τις επιθυμίες των ε, ενδιαφερομένων μέρων. Άλλοι ευρωβουλευτέ αναφέρθηκαν στη σημασία της βιοποικιλότητας και του κλίματος και πρότεινε μεγαλύτερη χρηματοδότηση να προέρχεται από την κοινή γεωργική πολιτική. Αναφέρθηκε και άλλες φορές αυτή η διασύνδεση μεταξύ της κοινή γεωργικής πολιτικής και της στρατηγικής για την βιοπικιλότητα. Και εδώ θα ήθελα να πω, το είπε ο κ. Γκερμπράντι, ρώτησε αν το στηρίζει πλήρω αυτό ο Επίτροπος Χόγκαν. Ήταν ομόφωνη η θέσπιση αυτού του σχεδίου δράση και από τον έλεγχο καταλληλότητα κατά κύριο λόγο προέκυψε ότι πρέπει να υπάρξει καλύτερη ε, αλληλεπίδραση με την κοινή γεωργική πολιτική. Το σχέδιο δράσης θα ενισχύσει την αλληλεπίδραση αυτή. Πρέπει να γίνει καλύτερη χρήση των πόρων, πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη ε, προσέγγιση. Όμως ε, το σχέδιο δράσης δεν μπορεί να αντιμετωπίσει όλους τους περιορισμούς της ε, ΚΑΠΑΓΑΜΑΠΗ ε, που θα συζητηθεί βεβαίως για η αναθεώρησή της στη συνέχεια της χρονιάς. Η κυρία Γκροστέτ, ξέρετε, μάλλον εσείς μόλις αναφέρατε ότι αποτελεί αυτή αποτελούν θεμελιολήθο αυτές οι δύο οδηγίες. Και σας ευχαριστώ για αυτή την παρατήρηση. Μιλήσετε για πολύ σημαντικά ζητήματα. Ποια είναι, ποιο είναι το κόστος και τα ωφέλη. Βεβαίως και τα ωφέλη Αυτά υπερβαίνουν μόνο την ε, απλή ε, συνεκτίμηση του κόστους και του ωφέλους ε, της βιοπικιλότητας. Και μιλήσατε και εσείς συγκεκριμένα για την ευελιξία σε ό,τι αφορά τον λύκο, όπου εφαρμόζονται οι οδηγίες πολύ περιοριστικά. Και εγώ θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχει τρόπος, υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις που επιλύουν τέτοια προβλήματα που αφορούν συγκεκριμένα είδη. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούν, μπορεί κανείς να λάβει συγκεκριμένα μέτρα, όμως όλα αυτά βάσει ε, ενός συγκεκριμένου διαχειριστικού σχεδίου και σε μια επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να εργαστούμε από κοινού και μαζί με την τοπική κοινωνία. Υπάρχουν πολλές ε, σε πολλές περιοχές τη Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν περιπτώσεις όπου τελικά βρίσκουμε μία ισορροπημένη λύση και βεβαίω ε, σας διαβεβαιώ για την ε, βούλησή μας να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια. Ήρθαν και εκπρόσωποι της Επιτροπής των Περιφερειών από τη Γαλλία, μου μίλησαν και νομίζω ότι και με τον guidance θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια. Έφυγε ο κ. Γεμπράντη, κρίμα γιατί ήθελα να τον ευχαριστήσω για την παρέμβασή του υπέρ της βιοπικιλότητας. Θα ήθελα να τον διαβεβαιώσω ότι ακριβώς μας απασχολεί η ευρύτερη εικόνα και όχι τα επιμέρους περιστατικά. Μίλησε για το χρονοδιάγραμμα, τέλη Απριλίου όπως προανέφερα, ανάγκες χρηματοδότησης των μελών. Θα έχουμε τη δυνατότητα να, εντοπίσουμε τις ανάγκες και τρίτον απάντησα ήδη για την κοινή γεωργική πολιτική η κυρία Γκέρλινγκ ανέφερε την αξία που ε, προσδίδουν οι πολίτες στην βιοπικιλότητα, Πράγματι κάποιες φορές είναι λυπής και γι' αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε τη διαβούλευση με τα ενδιαφερμένα Μέρη. Κυρία Πιατικά, έναν μίλησε για τα κάτι μελη Λοιπόν, αν υπάρχουν πράγματα τα οποία έχω ξεχάσει, βεβαίως και να είμαι, είμαι στη διάθεσή σας να τα συζητήσουμε και διμερώς με τους ευρωβουλευτές. Κλείνοντας, να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι με αυτό το σχέδιο δράσης μπορούμε πραγματικά να επιφέρουμε βελτιώσεις, αν εργαστούμε από κοινού με τα κράτη-μέλη, με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τοπικές περιφερειακές αρχές, γιατί η βιοποικιλότητα αφορά τους πάντες. Και είναι ένας από τους τομείς όπου βλέπουμε τον αντίκτυπο του ενωσιακού δικαίου και ε, την ευθύνη που βαρύνει και εμάς ε, και τους ε, ψηφοφόρους μας σας μάλλον. Είμαστε ε, πεπισμένοι να βρούμε λύσεις, ε, δεν ε, θέλουμε να βρούμε ιδιαίτερα περιοριστικά πλαίσια που δεν μας επιτρέπουν να κάνουν τίποτα, αντιθέτω, όμως κλείνοντας πιο θετικά, αυτό το θέμα, αυτός ο φάκελος μας δίνει μια τρομερή ευκαιρία να αποκαταστήσουμε τις σχέσεις μας με τους πολίτες μας, να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη, να τους δείξουμε έναν τομέα πολιτικής όπου υπάρχει πραγματική βελτίωση σε ό,τι φορά την προστασία του περιβάλλοντος, τη βιοπικιλότητα αλλά και την οικονομία. με την προώθηση βιώσιμων πρακτικών. Και τελικά έτσι δίνουμε πολύ καλά αυτά αποτελέσματα στους πολίτες μας. Ας ελπίσουμε ότι θα καταλήξουμε σε ένα πολύ καλό ε, σχέδιο δράσης, το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε μαζί σας, να το υλοποιήσουμε να γιορτάσουμε την επέτειο ε, του Natura 2000 και επιτέλους να ανασχέσουμε αυτή την ε, ε, πτωτική πορεία της βιοποικιλότητας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Γενική Διευθυντά. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Προσμένουμε την 25η Μαΐου λοιπόν για να γιορτάσουμε, μάλλον την 21η Μαΐου, λέει πρόεδρος, για να γιορτάσουμε λοιπόν την επέτειο αυτή της των δύο Τώρα, σας ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι για την υπομονή σας. Περιμέναμε μέχρι τώρα για να συζητήσουμε το τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Την εφαρμογή δηλαδή της οδηγίας 2004 κάθετος 35 σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας εισηγητής είναι ο κύριος Γιάβορ και θα του δώσω αμέσω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφε, η οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη είναι βασική ε, νομοθεσία για την δημιουργία περιβαλλοντικής ευθύνης χρησιμοποιώντας την αρχή του ορυπαίνων πληρώνει και ε, για να υπάρχουν μέτρα αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημίας. Πρόσφατα έγινε μία ε, επανεξέταση της οδηγίας στα πλαίσια του Ριφίτ για να δούμε αν είναι ακόμα κατάλληλη και η αρχική ε, εικόνα που αποκομίσαμε μετά από την ε, υποβολή θέσεων των κρατών μελών δημοσιεύτηκε πρόσφατα. Σε ό,τι αφορά τη δουλειά μας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή Περιβάλλοντος θα γνωμοδοτήσει σε μια έκθεση της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων για την έκθεση εφαρμογής της ε, οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη είναι συνδεδεμένη επιτροπή υπό τον κανόνα 54. Τώρα, ε, τα ευρήματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει ότι παρά τις βελτιώσεις που έχουν γίνει, η οδηγία έχει, ε, χαρακτηρίζεται ως όχι τόσο αποτελεσματική. Υπάρχουν μάλιστα τεράστιες διαφορές από κράτος μέλος σε κράτες μέλος και υπάρχει ένα σύνολο, ένα κολάζ ε, νομοθεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες όλες βρίσκονται κάτω από, την, ε, το ίδιο πλαίσιο. Αυτό κινδυνεύει να υπονομεύσει τα κοινά πρότυπα και ε, κινδυνεύουν με οικολογική καταστροφή πάρα πολλά μέρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η γνωμοδότησή μου νομίζω καθιστά σαφέ ότι χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε ε, με συστημικό τρόπο τις ε, προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας και να εξετάσουμε το μέλλον της οδηγία αυτής στα πλαίσια του refit. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις ε, προκλήσεις μας εν ώψη του πολιετούς προγράμματος εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δίνει έμφαση στην παροχή ε, κατάλληλης και παρκούς στήριξης στα κρατη Πέραν αυτών, πιστεύω πως ε, μία αναθεώρηση θα μας επιτρέψει να διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογή και ε, της ε, οδηγίας και να αναλυφθεί ευθύνη από τους ε, από τους ε, αρμόδιους φορείς και να γίνουν πιο αυστηρά τα κριτήρια. Θα ήθελα τέλος να κάνω έκκληση στην Επιτροπή να επιβάλλει κυρώσεις ε, για την έλλειψη ανάληψης ευθύνης ε, σε θέματα που έχουν να κάνουν με τη δημόσια υγεία. Επιπλέον, κάτι που θεωρώ πολύ σημαντικό είναι πως υπάρχει ανάγκη να επανεξετάσουμε το, τη χρηματοδότηση των ε, μέσων εφαρμογή οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη. Αυτό ίσω χρειαστεί αλλαγή των ανώτατων ορίων για την ε, ασφάλεια, για του ε, χειριστέ των προγραμμάτων. Θα μπορούσαμε επίση να εξετάσουμε τον δεχόμενο δημιουργία ενό Ευρωπαϊκού Ταμείου για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και τη δημιουργία πρόσθετων μέτρων για την αντιμετώπιση καταστροφών μεγάλης κλίμακας. Επίσης, η κατάλληλη ε, παρακολούθηση, ο κατάλληλος έλεγχος των αρμόδιων αρχών, είναι πάρα, ε, αρχών εφαρμογής είναι πάρα πολύ σημαντικός. Αυτό το είδαμε και στην προηγούμενη κουβέντα που είχαμε για τη συζήτηση για τους φυσικούς οικοτόπους, αλλά ε, βλέπουμε πόσο σημαντικό λοιπόν είναι ε, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει ακόμα περισσότερες δυνατότητες ελέγχου και επικοινωνίας με τους εθνικούς αρμόδιους φορείς. Γι' αυτό λοιπόν θα ακούσω τα σχόλια και τις προτάσεις σας με μεγάλη χαρά και ελπίζω να λάβω τις τροπολογίες σας. Η καταληκτική ημερομηνία της τροπολογίας είναι 25 Απριλίου και να πω πως είμαι σίγουρος πως το σχέδιο γνωμοδότησης ε, που έχω ε, ετοιμάσει μπορεί να βελτιωθεί πάρα πολύ από τις δικές σας προτάσεις. Και επιτρέψτε μου ένα τελευταίο σχόλιο. Υπάρχει μια δημόσια ακρόαση για το θέμα αυτό που θα γίνει το βράδυ της 11 η Απριλίου. Είναι μια κοινή ακρόαση με τη συμμετοχή της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων και εκεί θα έχετε τη δυνατότητα να ε, μάθετε περισσότερα. Θα υπάρχουν εμπειρογνώμονε εκτό Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σίγουρα πιστεύω θα είναι μια πολύ επικοδομητική συνεδρίαση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιάβολ. Η κυρία Πιετικάινεν έχει ε, το ρόλο της κοιόδουσης συζυγήτριας για την γνωμοδότηση αυτή, εκ μέρους του ΕΛΚ και θα σας δώσω το λόγο, παρακαλώ να μείνετε στα δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και τον εισηγητή η νομοθεσία για την περιβαλλοντική ευθύνη είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λήθους ε, τη ε, θεσμικής μας αντιμετώπισης ε, περιβάλλοντος. Πολλές φορές βλέπουμε ότι κάποιος την πληρώνει, είτε είναι οι μελλοντικέ γενιές, είτε είναι οι αγρότες και βλέπουμε όμως ότι υπάρχουν και κάποιοι που επωφελούνται δωρεάν, χωρίς ανταπόδοση. Χρειάζεται επομένω να αναλυφθεί ευθύνη από όσου αποφελούνται του περιβάλλοντο και τη χρήση τη γη. Υπάρχει νομοθεσία, αυτό το έχουμε δει. Υπάρχουν όμω ε, τρία κύρια χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να έχουμε υπόψη μα ε, σε οτιδήποτε κάνουμε εδώ στο Κοινοβούλιο. Πρώτον, ποιο είναι το εύρο τη νομοθεσία, ποιε είναι οι δράσει που συμπεριλαμβάνει η πρόταση τη Επιτροπή και ποιε είναι οι νέε προτάσει. Ε, υπάρχει πρόταση να συμπεριληφθούν όλες οι οικονομικές δραστηριότητες και οι εσκεμμένες και μη εσκεμμένες δράσεις που έχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ε, και επίσης η εξόριξη είναι ένα πολύ καυτό ζήτημα σε πολλά κρατημέλη. Έπειτα, η ερμηνεία της νομοθεσίας, ε, τι σημαίνει η ευθύνη, ποιος πληρώνει, πόσο πληρώνει. Εδώ πιστεύω πως είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές από κράτος σε κράτος και έπειτα υπάρχει και το βάρος της απόδειξης. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ξέρουμε ακριβώς ε, πόσο κοστίζει το κόστος. Και έπειτα δεν ξέρω πώς ακριβώς η φύση μπορεί να επανέλθει από την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει τώρα και αν δεν μπορεί να επανέλθει, τι μπορούμε να κάνουμε, πώς θα βρούμε επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του τουρισμού, αγρότες και τα λοιπά που θα χρησιμοποιήσουν στο μέλλον τη γη όταν η ποιότητα της γης έχει εκφυλιστεί. Και έπειτα ε, στα πλαίσια της αναθεώρησης πιστεύω πως πρέπει να δώσουμε βάρος στις κυρώσεις, στο κόστος και ε, στις αποσμιώσεις. Κάτι που βλέπω πως λείπει από την οδηγία έτσι όπως είναι τώρα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και μίλησα δύο λεπτά, λέει κυρία Κάινεν. Το πρόσεξα, λέει πρόεδρο. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι σχεδόν ηγετής των σοσιαλδημοκρατών, Όμω θα τον εκπροσωπήσει η κυρία Ντάλι και έχετε το λόγο. Σα ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους του Νίκου Ανδρουλάκη για την απουσία του σήμερα και να ευχαριστήσω τον κύριο Γιάβορ για την ε, δουλειά που έκανε ως εισηγητής αυτής της γνωμοδότησης. Η ομάδα μας συμφωνεί με όλες τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις που βρίσκονται στη γνωμοδότηση Θεωρούμε πως η περιβαλλοντική ευθύνη και η οδηγία αυτή έχει επηρεάσει ε, την ε, κατάσταση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε όλη την Ευρώπη. Ωστόσο, όπως ήδη ακούσαμε, πολλά θέματα ακόμα είναι ε, στα χέρια των κρατών μελών. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε υπέρ μιας αναθεώρησης το συντομότερο δυνατόν της οδηγίας αυτής, έτσι ώστε να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο αναρμόνησης και θεωρούμε επίσης πως χρειάζονται αυστηροί κανόνες ε, περί ευθύνη για όλες τις περιπτώσεις περιβαλλοντικής ζημίας, ιδιαίτερα ε, δεδομένη της πρόσφατη εμπειρία μας ε, με το σκάνδαλο των εκπομπών. Γι' αυτό θεωρούμε πως πρέπει να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής και να συμπεριλαμβάνει την, δημόσια υγεία και ε, τα υπόλοιπα που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα 3. Επίσης, ας ε, κοιτάξουμε ξανά τη, το να δημιουργήσουμε μία υποχρέωση για χρηματοδοτικά μέσα, για ενίσχυση των εφορέων και ας φροντίσουμε έτσι ώστε να εφαρμόζεται πάντα η αρχή του ορυπαίνων πληρώνει. Αυτά λοιπόν εκ μέρους του κύριου Ανδουλάκη. Να σας πω επίσης ότι με χαρά θα ε, παρευρεθεί στην ακρόαση με την Επιτροπή Γιούρη και θα ήθελα να ευχαριστήσει όλους τους κοιόδης εισηγητές και τους υπόλοιπους συναδέλφους. Ευχαριστώ. Ναι, για τον Απρίλη είχαμε την ακρόαση. Επόμενος σκιώδης. Η κυρία Γιάτα Βάκα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς τους συναδέλφους και τον κύριο Γιάβορ για το σχέδιο γνωμοδότησης. Εδώ βλέπω πως θίγονται ζητήματα τα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη ε, παρουσίασε τον περασμένο Απρίλιο ο ρηπαίνων πληρώνει είναι η βασική αρχή που πρέπει να ακολουθήσουμε και είναι κάτι το οποίο πιστεύω θα αποτελέσει το, το επίκεντρο των συζητήσεων στην επόμενη συνάντηση των σκιωδών εισηγητών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν διασφαλίσεις για όλους τους εμπλεκόμενους ε, φορείς, διότι όλοι γνωρίζουμε πως ε, υπάρχουν μεγάλες διαφορές από κράτος σε κράτος και πως η εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο δεν έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα, απέχει πόρο από αυτά, ιδιαίτερα σε ορισμένες χώρες. Πολλές φορές ε, γι' αυτό ευθύνονται οι, οικονομικοί, οι οικονομικές συνθήκες, η έλλειψη πόρων, αλλά πολλές φορές και η διαφθορά ή η έλλειψη ενδιαφέροντος. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους ορισμούς και τις, ε, ε, και τις ε, σχετικές διατάξεις, εδώ νομίζω πως υπάρχει περιθώριο λιγμών, αλλά αυτό είναι και το πρόβλημα. Μπορεί να οδηγηθούμε σε τεράστιες διαφορές στην εφαρμογή. Γι' αυτό χρειάζεται σαφήνεια και ξεκάθαρος προσανατολισμός. Δεν είμαι όμως σίγουρη για το αν θα ωφελήσει αυτό το νέο χρηματοδοτικό μέσο που αναφέρατε. Νομίζω πως εδώ ξεπερνάμε τα όρια και ξεπερνάμε και τα όρια της ε, χρηματοδότησης. Σίγουρα βέβαια χρειάζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού, όμως τώρα μια νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία δεν είμαι σίγουρος που μπορεί να ωφελήσει. Το θέμα είναι να λειτουργήσει το σύστημα που έχουμε ήδη στη διάθεσή μας. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι δεν λειτουργεί, όχι να δημιουργήσουμε άλλο. Μετά, υποχρεώσεις των κρατών μελών. Αυτό θέλει σκέψη. Είναι σίγουρα κάτι που πρέπει να εξετάσουμε. Ε, θέλω λοιπόν να ευχηθώ σε όλους καλή δουλειά. Γιατί η δουλειά δεν είναι μόνο στα κράτη-μέλη, αλλά πρέπει να κάνουμε και εμείς εδώ το δικό μας κομμάτι. Grazie, Ευχαριστώ κύριε Σποδοσύνη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να κάνουμε ένα πείραμα. Να μας πούν οι Ευρωπαίοι πολίτες τι άποψη έχουν για το ρηπαίνον πληρώνει. Εγώ είμαι βέβαιος ότι περισσότεροι θα έλεγαν ότι δεν υπάρχει αυτή η αρχή. Ένα μικρό κομμάτι θα έλεγαν ότι ξέρουν ότι υπάρχει και ότι εφαρμόζεται, αλλά με δυσκολίες και το υπόλοιπο πείμα θα έλεγε ότι είναι δύσκολο να εντοπίσουμε τους υπεύθυνου και να τους τιμωρήσουμε. Υπόθηκε εξάλλου ότι μόνο το 10, το 2010 καταγράψαμε την πλήρη μεταφορά της οδηγίας για την ευθύνη και με αποκλήσεις μεταξύ χωρών μελών. Και είχαμε χιλιάδες περιβαλλοντικέ υποθέσει από το 7 μέχρι το 10, όπου χώρε όπου η Ουγγαρία ή η Πολωνία κατέγραψαν το 86% αυτών των περιπτώσεων. Ενώ σε κάποιε χώρε 10, δεν είχαμε κανένα, καμία υπόθεση. Για την Ιταλία, όπως λέει η Κομισιόν, εμείς έχουμε εφαρμόσουμε πιο επικτατικό, πιο ευρύ τρόπο την οδηγία από ό,τι χρειάζεται. Και έχουμε καταγράψει 17 περιπτώσεις 12 σε σχέση με καταβολές κονδυλίων και 5 για βλάβες. Φαίνεται λοιπόν ότι η Ιταλία τα πάει καλά σύμφωνα με την έκθεση της Κομισιόν. Όμως στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις έχει ξεκινήσει η διαδικασία ώστε να πληρώσουν αυτοί που είναι υπεύθυνοι. Όμω δυστυχώ η κατάσταση είναι τελείω διαφορετική. Γιατί όλοι οι Ιταλοί πολίτε γνωρίζουν τι βλάβε τι περιβαλλοντικέ που λαμβάνουν χώρα στη χώρα μα. Ε, στην Νότια Ιταλία, στο Τάραντο, η απόρριψη των πυρηνικών αποβλήτων στη θάλασσα, παράνομε χωματερές κλπ. Οπότε εμεί αναρωτιόμαστε τι έγινε με αυτή την οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη. Ισχύει σε αυτές τι περιπτώσεις που ανέφερα. Γιατί η αρχή στην Ιταλία είναι ότι ο πληρώνων, ο συγγνώμη, δεν πληρώνει. Ευχαριστώ, λέει πρόεδρο. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Ζητάμε μια αναθεώρηση τις οδηγίες για την ε, περιβαλλοντική ευθύνη. Αυτό είναι κάτι παγκοσμίω πρωτοεμφανιζόμενο και μάλιστα έχουμε να κάνουμε θέματα τα οποία έχουν μορφή παγκοσμίου ρεκόρ. Εδώ έχουμε κάτι το οποίο έχει μορφή αστικής ευθύνης, αλλά βλέπουμε ότι αυτό δεν συνάδει με την περιβαλλοντική ευθύνη. Αυτό έχει να κάνει βέβαια με τα διακυβευόμενα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να εφαρμόσει ένα ενιαίο μοντέλο ευθύνη σε περίπτωση περιβαλλοντική βλάβη. Βεβαίω μπορεί να προωθήσει κάποια μοντέλα ευθύνη, σύμφωνα βέβαια και με την νομοθεσία τη Ένωση σε σχέση με την ε, προστασία τη ανθρώπινη ζωή και του περιβάλλοντο. Θα πρέπει λοιπόν να πλαισιώσουμε τις αποκλήσεις που έχουν να κάνουν με τις άδειες από τις ε, άδειες που έχουν να κάνουν με την, με την ανάπτυξη. Η αρχή του ερπαίνου πληρώνει δεν θα πρέπει να παρακαμφθεί, γιατί έχουμε να κάνουμε μεγάλες αποκλήσεις όσον αφορά τις βλάβες. Εξάλλου, όταν έχουμε έναν υπεύθυνο φορέα, ο οποίος δεν μπορεί να πληρώσει τις κυρώσεις που απαιτούνται, μπορεί κανείς να προστρέξει στην ε, χώρα μέλος, αλλά χωρίς να, υπάρχουν, να υπάρξουν, χωρίς να πρέπει να υπάρχουν επιβολές στις φορολογούμενους. Θα πρέπει επίση να δούμε τι γίνεται με τη χρηματοδότηση αυτών των αποκαταστάσεων. Για, την, για το όριο ευθύνη τώρα που ποικίλει, θα πρέπει να κάνουμε μια πρόληψη των βλαβών. Δηλαδή θα πρέπει να αποφασίσουμε ποιο θα πληρώσει σε σχέση με τι υποχρεωτικέ χρηματικέ εγγύησει. Αντί να δημιουργήσουμε λοιπόν ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο τη Ένωση για την αποκατάσταση, νομίζω ότι το διεθνέ πλαίσιο είναι πολύ πιο λειτουργικό και θα πρέπει να το δούμε. Εξάλλου αυτό θα μας επέτρεπε να έχουμε μια πιο συνεπή δράση όσον αφορά τις ε, μεγάλες διοσυνοριακές διεθνικές βλάβες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Λέκη Πρόεδρος. Τώρα ο κ. Δετζένι από την Κομισιόν. Καλησπέρα Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Και ευχαριστώ που θέσατε αυτό το σημείο στην ημερήσια διάταξη. Χαίρομαι πολύ που εξετάζετε τη δουλειά που έχουμε κάνει στα πλαίσια αυτής της οδηγίας. Και θα θέλαμε να ακούσουμε τις απόψεις σας και να λάβουμε την συμβολή σας για το πώς θα προχωρήσουμε. Να ευχαριστήσω και τον εισηγητή, τον κύριο Γιάβορ, με το οποίο είμαστε σε επαφή εδώ και χρόνια. Είναι σημαντικό για μας, αφενός, να μοιραστούμε την ανάλυση που κάνουμε στα πλαίσια της έκθεσης αξιολόγησης. Αλλά βέβαια να συζητήσουμε και μαζί και να σας ακούσουμε για το ποιες είναι οι καλύτερες δυνατές λύσεις για να σημειώσουμε πρόεδρο. Να συνοψίσω σύντομα τι έχουμε κάνει και τι πρόοδος έχει σημειωθεί από την εθέντηση της έκθεσης. Πρόοδο και τι σχεδιάσουμε να κάνουμε. Όπως είπατε κι εσείς, έχουμε δημοσιεύσει μία έκθεση. Αυτό έγινε πέρσι, στα πλαίσια της αξιολόγησης. Τονίσατε και προγραμμίσατε διάφορα ζητήματα και επιμέρου θέματα. Θέλω όμως να σας πω ότι το ότι υπάρχει οδηγία σχετικά με την ευθύνη έχει επιτρέψει τη σύγκληση των μοντέλων ευθύνε στην Ευρώπη. Βεβαίω κάποιε χώρε ήδη είχαν κάποια πλαίσια ευθύνη, άλλε δεν είχαν τίποτα. Και γι' αυτό ακριβώ καταλήξαμε στην οδηγία. Πρέπει λοιπόν να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει πρόοδο σημαντική σε κάποιε χώρε μέλη σχετικά με την εφαρμογή τη οδηγία. Αναφέρθηκε όμω ότι κάποιε ε, χώρε μέλη δεν έχουν αναφέρει καμία υπόθεση περιβαλλοντική. Ίσως λοιπόν να πει κανείς ότι δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε αυτό το εργαλείο γιατί τα εθνικά μας εργαλεία μας επιτρέπουν να έχουμε τα αποτελέσματα. Και εδώ ακριβώς νομίζω θα πρέπει να επικεντρωθούμε ώστε να μπορέσουμε να αποδείξουμε ότι πετυχαίνουμε τους συνολικούς στόχους που έχει θέσει η οδηγία. Είτε μέσω εργαλείων ενωσιακών, είτε μέσω συμπληρωματικών εθνικών εργαλείων. Και αυτό προσπαθήσαμε να το εξετάσουμε στην αξιολόγησή μας. Γι' αυτό ακριβώς λοιπόν προτείναμε διάφορες δράσεις στην έκθεσή μας και ήδη έχουμε ξεκινήσει τη δουλειά σε αυτές τις δράσεις. Αφενός λοιπόν, όπως είπατε και πολλοί από εσά, σίγουρα θα πρέπει να θεγραμμίσουμε τις ε, δράσεις εφαρμογής. Έχουμε κάποια καλά παραδείγματα και θα θέλαμε σε συνεργασία με τις χώρες μέλη και όπως στην οδηγία για τους βιοτόπους να πάμε σε μια αντίστοιχη εφαρμογή με παρόμοιε δράσει και εξετάσουμε αυτή τη στιγμή ποιε είναι οι καλύτερε δυνατέ πρακτικές, κατευθύνσει γραμμές κλπ. Δεύτερον, τα αποδεικτικά στοιχεία. Θεωρούμε ότι αν δεν ξέρουμε συγκεκριμένα τι έχει συμβεί σε διάφορε περιβαλλοντικές υποθέσει ποια είναι η κατάσταση, και για ποιο λόγο δεν εφαρμόζεται η οδηγία, τότε θα πρέπει να γνωρίζουμε τι γίνεται ακριβώ, το οποίο αποτελεί μια προπόθεση για οποιαδήποτε συζήτηση για το ίδιο το εργαλείο. Γι' αυτό ακριβώ το λόγο με χαρά σα ενημερώνω ότι σε μια πρόσφατη συνάντηση εμπειρογνωμόνων των Εθνικών Αρχών μπορέσαμε να πείσουμε του εμπειρογνώμενου των χωρών μελών για τη σκοπιμότητα του πολιετούς προγράμματος εργασίας το οποίο θα δημοσιευθεί αυτή η εβδομάδα την ερχόμενη κάτι το οποίο θεωρούμε ως ένα δικό χάρτη απτό σε σχέση με την εφαρμογή των δράσεων που θεωρούμε ότι είναι σημαντικές για να βελτιώσουμε την εφαρμογή. Τώρα, για την ασφάλεια τη δημοσιονομική θεωρούμε ότι ήδη υπάρχουν κάποια εργαλεία σε κάποιες χώρες και συστήματα, άλλες χώρες δεν διαθέτουν τέτοια συστήματα και έχουν μείνει πίσω. Ξέρουμε όμως ότι αυτό το θέμα είναι δύσκολο και το είδαμε σε διάφορες εκθέσεις. Προσπαθούμε λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο εμπειρογνωμόνων στις διάφορες χώρες μέλη για να δούμε ακριβώς πώς θα μπορούσαμε περαιτέρω να ενισχύσουμε την εφαρμογή <coughs> της νησονομικής ασφάλειας σε όλες τις χώρες μέλη. Και γι' αυτό ακριβώς πρόσφατα δημοσιεύσαμε την επιθεώρηση όπου εκεί ακριβώς αναφερόμαστε συγκεκριμένα σε χώρες μέλη όπου θα πρέπει να βελτιωθεί η εφαρμογή και υποβάλλουμε αντίστοιχε προτάσεις για επιμέρους ζητήματα. Και αναφέρουμε ακριβώς και τις χώρες μέλη όπου χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια για την δημοσιονομική ασφάλεια. Αυτά είναι αναπόσπαστο κομμάτι όλων των συνολικών προσπαθειών για τη βελτίωση της εφαρμογής ώστε να πετύχουμε τους συνολικούς στόχους της οδηγίας σε όλες τις μέλη. Καταλήγοντας να σας πω ότι για μας δεν είναι ακόμα η κατάλληλη στιγμή, δεν έχει έρθει για την αθεώρηση της οδηγίας. Θεωρούμε ότι μπορούμε με τα εργαλεία που έχουμε να πετύχουμε περισσότερα. Κάποια στοιχεία που προτείνει στην έκθεση του κ. Γιάβορ ήδη μπορούμε να τα εφαρμόσουμε στα πλαίσια της υπάρχουσας οδηγίας, απλά και πρέπει να ασφαλίσουμε ότι αυτό γίνεται, αλλά κατά μεριά δεν είμαστε και κάθετα αντίθετοι άκουσα τη συζήτηση, άκουσα τις ε, προτάσεις. Είπε ο κ. Γιάβορ κάτι για πρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προοπτικέ. Θέλουμε λοιπόν να συμμετάσχουμε στι ακροάσει σα και να συνεργαστούμε μαζί σας, όπως και σε, με άλλε επιτροπέ του Κοινοβουλίου, ώστε να έχουμε μια καλή βάση διαλόγου για το πώς θα αναπτυχθεί αυτό το εργαλείο βράχη πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα στην οδηγία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Λάκη Πρόεδρος. Ο συγγετής μας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους σας για τις παρατηρήσεις. Νομίζω ότι υπάρχει συνένεση μπορούμε να συμφωνήσουμε πάνω σε πολλά ζητήματα, οπότε θα έχουμε μια οικοδομητική συνεργασία νομίζω. Υπάρχουν και κάποια άλλα ενδιαφέροντα ζητήματα, όπως είναι η δημοσιονομική ασφάλεια. Δεν θα ξεκινήσω τώρα συζήτηση. Ευχαριστώ να κάνουμε λεπτομερή συζήτηση όταν το αντίστοιχο σύστημα θα υπάρχει γιατί αυτή τη στιγμή υπό την τωρινή μορφή της οδηγίας δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Πρέπει λοιπόν στα πλαίσια της οδηγίας να συγκροτήσουμε ένα αποτελεσματικό σύστημα αυτού του είδους. Και αυτό θα πρέπει να γίνει πανευρωπαϊκά ώστε ο περιβαλλοντικός κίνδυνος να αφορά εξίσου όλες τις χώρες και τους πολίτες. Αλλά και για να υπάρχει και μια δυνατότητα για τις ε, επιχειρήσεις και για την οικονομία να αναλάβει τις δικές της ευθύνες. Γιατί νομίζω ότι πολλές περιβαλλοντικές ε, βλάβες έχουν διασυνοριακή φύση. Οπότε Πρέπει να έχουμε ένα ευρωπαϊκό σύστημα, επειδή ακριβώς έχουμε διαφορετικά καθεστώτα σε διάφορες χώρες και αυτό δημιουργεί προβλήματα. Αλλά βεβαίω προσβλέπω σε περαιτέρω συζήτηση με τους κοιόδης εισηγητές και αναμένω βέβαια και τις δικές σας συμβολές μέσω των τροπολογιών. Και πιστεύω ότι τελικά θα εκπονήσουμε κάτι το οποίο θα είναι αποδεκτό από την Επιτροπή και θα είναι καλό. Ευχαριστώ να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε αυτή την κοινή ακρόαση με τη Γιούρη στις 11 του Απρίλη και έχουμε μία προθεσμία τροπολογιών 8 Ιούνιου. 28 Απρίλη διορθώνει τώρα η Πρόεδρος. 28 Απρίλη, 11 ώρα το πρωί. Άλλαξε. Επόμενη συνεδρίαση, 10 του Απρίλη. Ευχαριστώ. Τέλος συνεδρίωση. Γεια σας.